On test. Λοιπόν, να κάνουμε μια δοκιμή. Ε, άρχεται η ψηφοφορία. Κύριε Μπουλόν. <laughs> Bien, Πέρα ψηφοφορίες. Λοιπόν, δυο. Il en manque un. Μία ψήφος λείπει. Eh ben, c'est bon. Dax, Tout le monde voté Εντάξει. 23. Voilà, tout le monde a voté en faveur du vote. Έρχεται και ο κύριος Κασμάρεκ, οπότε αρχίζουμε με την έκθεση για το, τις ε, τοπικές ε, ε, αρχές ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η πρώτη παράγραφος συμβαστική λύση 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 2 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική λύση 2 υπέρ κατά αποχές η 16 καταπίπτει 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 19 υπέρ κατά αποχές Ας ελέγξουμε την τροπολογία 19. Ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική, συμβαστική 3. 3 και Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 23. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 26 σε δύο μέρη πρώτο μέρος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο μέρος υπέρ κατά αποχές ας το ελέγξουμε για το δεύτερο τμήμα της 26 πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται 7. Παράγραφος 7. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 28. Υπέρ κατά εγκρίνεται. Ε, συμβαστική λύση 4. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 30. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 31. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τώρα 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 51 τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 52 έως 54 όλες μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 55 και 58 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 59 σε τρία μέρη, πρώτο μέρος υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, δεύτερο μέρος υπέρ, κατά, αποχές, α, Ας το επαληθεύσουμε. Ψηφίζουμε για το δεύτερο μέρος, παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τρίτο μέρος, υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε. Ψηφίστε. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 60 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 61 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Πάμε τώρα... Σε αιτιολογικές σκέψεις 3 έως 5 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται, τροπολογία 6. Για να ψηφίσουμε Ψηφίστε για την έξι. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 7 έως 9 τροπολογίες υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Αναφορές. Να τις πάρουμε όλες μαζί και τις τέσσερις υπέρ υπέρ κατά εγκρίνονται κατά εγκρίνονται τελικώς είδατε πάω πιο γρήγορα τελική ψηφοφορία διανατάσεως χειρός υπέρ κατά αποχές όχι πρέπει να το κάνουμε ηλεκτρονικά ψηφίστε πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. Είδατε καλά το μάντεψα. Και δει με ομοφωνία. Συγχαρητήρια. Oui, Γυναίκες με αναπηρία. Μία και μόνη τροπολογία υπάρχει. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τελική ψήφος υπέρ, κατά, αποχή εγκρίνεται. Ψηφοφορία ηλεκτρονική. Ψηφίστε. Εγκρίνεται με ομοφωνία. Προχωρούμε για την περιοχή του Σαχέλα peut faire bloc Bloc, oui, oui. Je vous propose. Oui, oui, oui. Je vous propose en bloc l'amendement. Προτείνω τι τροπολογίε 1 έω 7, όλε. μέχρι την 5, 1 έω 5 λοιπόν. Ποιο είναι υπέρ, κατά, αποχέ εγκρίνονται. 6 υπέρ, κατά. Α το ελέγξουμε για την τροπολογία 6, ψηφίστε. Πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται. Τροπολογία 7 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 8 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 9 σε δύο μέρη. Πρώτο μέρος υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος υπέρ. Κατά αποχές. Για να το ελέγξουμε. Ψηφίστε ηλεκτρονικά. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Τροπολογία 10, 11, 12. Τροπολογίες μέχρι το 16, μέχρι 17. Όχι 16. Ωραία, 10 έως 16. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Τροπολογία 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 18. Υπέρ. Κατά. Αποχές... Α, να το ελέγξουμε τροπολογία 18 πέρας εγκρίνεται τροπολογία 19 μέχρι 25 19-25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τελική ψηφός υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ηλεκτρονική ψηφοφορία ψηφίστε πέρας εγκρίνεται με ομοφωνία. Επόμενη τώρα ε, ψηφοφορία ο κύριος Σβένσον. Ah Συγγνώμη δεν είχα προσέξει. Μετά από την προφορική ερώτηση έχω τρεις τροπολογίες ομαδών και για τις τρεις ποιοι είναι υπέρ λοιπόν. Κοιτάξτε ο κύριος Κάσμαν δεν μας παρακολουθεί. Ένα λεπτό λέει ο κύριος Λάστρα. La, la Για τις διακρίσεις. 273 με 278. έπεται του ψηφίσματος κανονικά. Υπάρχουν τρεις τροπολογίες εν πάση περιπτώσει. Δεν το έχετε. Okay. Λοιπόν και για τις τρεις ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές δεκτές. Τελική ψήφος ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές δεκτές. Ηλεκτρονική ψήφος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορίες. Δεκτή ομόφωνα. Τώρα ερχόμαστε στο ψήφισμα. Σας προτείνω πάλι ομαδών από την 8 μέχρι τη 12. Όχι. 8 και 9 τότε μόνο. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτές. 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 11 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Προφορική τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 13. Σε δύο τμήματα. Α, όχι, έχει καταπέσει 13, ξεχάστε το. 14, 15 και 16. Μαζί λοιπόν, όχι, όχι, 14 πρώτα, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή, 15 ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή, 16 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Πρώτη παύλα υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή, Τροπολογία 3. Υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Προφορική 1. Υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 5. Τροπολογία 5 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές δεκτό. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 6. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 7. Υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Τροπολογία 1 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Τελική ψήφος υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Ηλεκτρονικός έλεγχος, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Ομόφωνα δεκτό. Τι ωραία που τα λέμε, λέει η πρόεδρος. Επόμενη έκθεση, έκθεση Μίτσελ, τροπολογία 1 και 2, μαζί, και είναι υπέρ κατά, αποχές, δεκτή. Τελική ψήφος, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Ομόφωνα δεκτή. έκθεση του κυρίου Πόγκα. Δεν υπάρχει τροπολογία, είναι τόσο τέλεια η έκθεση Πόγκα. Μπράβο κύριε Πόγκα, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Πέραση ψηφοφορίας. Ομόφωνα. Α, υπάρχει μία αποχή. Λάθος, λάθος, λάθος. Ομόφωνα λοιπόν. Έκθεση Κάσμαρεκ. Έχουμε μία τροπολογία, την τροπολογία 1. Ευχαριστώ. Κατά. Αποχές, απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την Κάτσμαρεκ. Πέραστη ψηφοφορία. ψηφοφορίας. Δεκτή. Τελειώσαμε λοιπόν με τις ψηφοφορίες. Mais il n'y a pas un deuxième vote là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 Συνάδελφοι, περνάμε τώρα στην παρουσίαση της εκθέσεως νομοθετικής προτάσεως της Ευρωπαϊκής που μαζί της Ευρωπαϊκής Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλουμε σύμφωνα με το 225 τη συνθήκη σχετικά με τον συντονισμό των δανειστών ε, στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για την πρωτοβουλία του συναδέλφου Γκέι Μίτσελ είναι αποτέλεσμα μιας μελέτης που ζήτησε να υπάρξει η Επιτροπή μας για το κόστος του μη συντονισμού στον τομέα της αναπτυξιακής βοήθειας. Στόχος της νομοθετικής αυτής πρωτοβουλίας είναι να καταθέσει μια νομοθετική πρόταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ενισχύσει το συντονισμό των αναπτυξιακών πολιτικών των κρατών μελών. Θα έχουμε την δυνατότητα να ακούσουμε επίσης και ε, την άποψη της Κομισιόν και της Υπηρεσίας Εξωτερικών ε, Σχέσεων. Πρώτος λοιπόν ο μιλητής, ο εισηγητής μας, ο κύριος Μίτσελ. Κοιτάξτε, έχουμε ένα μικρό θέμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει φτάσει ακόμα, γι' αυτό παρακαλώ μη βιάζεστε. Δεν χρειάζεται να βιάζεστε κύριε Μίτσελ, σιγά σιγά. Ευχαριστώ συνάδελφοι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τους Κιώδης ε, γιατί με θάρρυναν, με υποστήριξαν ε, ε, διότι για να προσεγγίσουμε σωστά το ζήτημα, όντω πρέπει να πούμε σε κάποιο επίπεδο λεπτομέρειε, αλλά νομίζω ότι όλοι συμφωνήσαμε ότι χρειάζεται καλύτερο συντονισμό, κυρίω αυτού του χαλεπού καιρού που ζούμε και ζητούμε από όλου να υποφέρουν. Ε, λόγω κρίση στα κράτη-μέλη. Τον Ιούνιο του 2013 έγινε μια παρουσίαση εδώ στην Επιτροπή Ανάπτυξης για μια μελέτη που έφερε τον τίτλο «Το κόστος τη μη Ευρώπη στην αναπτυξιακή πολιτική». Ε, σε αυτή τη μελέτη δράζεται και η έκθεσή μου ε, που φέρει τον τίτλο ε, «Συντονισμός των δωρητών της ΕΕ όσον αφορά την αναπτυξιακή βοήθεια. Λοιπόν, θα ήθελα να σας ε, παραπέμψω σε αυτή την έκθεση, σε αυτή τη μελέτη. Είναι πάρα πολύ καλή και έχει και άλλα στοιχεία πέρα από το κόστος της μη Ευρώπης. Λοιπόν, στην έκθεσή μου επαναλαμβάνω ότι 800 εκατομμύρια ευρώ μπορούμε να εξοικονομήσουμε ετησίως μειώνοντας ε, μόνο και μόνο το κόστος ε, συναλλαγών. Αν οι δωρητές συγκέντρωναν τις προσπάθειες που κάνουν σε λιγότερες χώρες και σε λιγότερες δραστηριότητες. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό λόγω χρηματοπιστωτικής κρίσης ε, και της αυξανόμενης πολιτικής ανησυχίας. Ε, δηλαδή όλοι θέλουν ε, να καταδείξουν ότι είναι αποτελεσματικές οι δαπάνες για τις οποίες δεσμευόμαστε. Ο στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά το 0,56 της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας μέχρι το 2010 ακόμη δεν έχει επιτευχθεί και έχουμε φτάσει στο 2013. Και δυστυχώς ε, κάθε χρόνο επαναλαμβάνουμε τα ίδια. Ε, υπάρχει μεγάλη πίεση, ασκείται ε, πίεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτού του πολιτικού εγχειρήματος, οπότε η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να καταδείξει ότι έχει προσθέμενη αξία η συνολική αυτή η δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι υποδεέστερο το ζήτημα, είναι ζήτημα ε, ζωής και θανάτου. 23.000 παιδιά παιδένουν κάθε μέρα. Παλιότερα βεβαίως ήταν 36.000 την ημέρα, καλά τα νέα, αλλά αυτά τα παιδιά, ε, τα 13.000 ζουν χάρη σε ακριβώς αυτές τις προσπάθειες ε, της αναπτυξιακής ε, βοήθειας. Ε, η παιδική θνησιμότητα είναι 68 της Χιλής. Στην Ιρλανδία μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο το ποσοστό ήταν 48 στα χίλια και τώρα έχουμε φτάσει στα χαμηλότερα ποσοστά. 68 της Χιλίας λοιπόν δεν είναι και πολύ άσχημο ποσοστό να συγκρίνουμε με το τι γινόταν μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο σε διάφορα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ίδιο μπορούμε να κάνουμε και σε τι αναπτυσσόμενες χώρες εάν ε, συνδυάσουμε τις προσπάθειές μας. Ε, έχουμε ηγηθεί διεθνών προσπαθειών για το συντονισμό ε, των προσπαθειών των δωρητών για την αναπτυξιακή βοήθεια. Δυστυχώς όμως η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτό το τομέα είναι μάλλον σε εθελούσια βάση και άρα δεν ικανοποιητικός ο συντονισμός. Έχει ανακύψει μια νέα ευκαιρία χάρη στη συνθήκη τη Λισαβόνα, διότι έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση νομική βάση που μπορεί να ενισχύσει τη συνοχή και την αποτελεσματικότητα τη εξωτερική τη δράση. Σα εκμεταλλευτούμε λοιπόν αυτό το νέο δεδομένο, αλλά με πυγμή και με επιδεξιότητα κυρίω. Αυτό είναι το μήνυμα το βασικό που περνάω μέσα στην έκθεσή μου. Ε, υπάρχουν δύο σημεία που μα εμποδίζουν στο να προχωρήσουμε και να επιτύχουμε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Κατακαιρματισμό και επικάλυψη αφενό και αφετέρου Συνοριακή έλλειψη συντονισμού. Και τα δύο προβλήματα τα πραγματεύεται η Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του κώδικα διοντολογία για τον επιμερισμό εργασία και παρότι έχουν ε, έχουν γίνει κάποια θετικά βήματα τα τελευταία έτη, ε, ο αυξανόμενο κόστος της αναπτυξιακής βοήθειας και αυτή η επιθυμία να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα με τα ίδια λιγότερα κονδύλια πάλι δημιουργεί, εξακολουθεί να δημιουργεί πρόβλημα για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και λόγω της μη δεσμευτικής ε, του εθελοντικού χαρακτήρα της δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την έλλειψη συντονισμού ε, δεν έχουμε εκμεταλλευτεί στο έπεκρον το δυναμικό που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να είναι πιο αποτελεσματική η αναπτυξιακή της βοήθεια βοήθεια και άρα χρειαζόμαστε ένα νέο όργανο συντονισμού που θα πάρει τη μορφή ενός κανονισμού. Ε, ποιες είναι οι συστάσεις λοιπόν που συμπεριλαμβάνονται στην έκθεσή μου. Για να επιτύχουμε το στόχο συστήνουμε έναν κανονισμό το οποίο το παιδί εφαρμογή θα προσφέρει και την πιο πρόσφορη λύση για αυτό το ζήτημα, δηλαδή πώς να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα τη επιδόση αναπτυξιακή βοήθεια. Πρόσφορο λέμε, μάλιστα. Εντάξει, κάποια πράγματα κάνουν τα κράτη-μέλη, κάποια άλλα τα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να συζητήσουμε τον ε, επιμερισμό. Ω προ τι αρχέ που πρέπει να προαγάγουμε και να υποστηρίζουμε, Έχουμε ένα κωδικοποιημένο σετ αρχών που έχουν ρόλο κλειδί για την αποτελεσματικότητα, εναρμόνιση, ευθυγράμμιση, διαφάνεια ε, και αμοιβή λογοδοσία καθώς και διαφοροποιημένη προσέγγιση. Ως προς τις ε, δράσεις που πρέπει να αναλυφθούν, η έκθεσή μου βασίζεται στο υφιστάμενο οπλοστάσιο, το πω έτσι, των πρωτοβουλειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που καθοδηγούν τα κράτη-μέλη αλλά και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, με στόχο την επίδειξη μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας. Ο Ευρωπαϊκός Κώδικα Διοντολογίας για την συμπληρωματικότητα και τον επιμερισμό ε, των καθηκόντων για την αναπτυξιακή βοήθεια θα πρέπει να υλοποιείται σε όλες τις ε, χώρες ε, όπου δραστηριοποιούμαστε ε, και χρειαζόμαστε μια συμφωνία πλαίσιο για να επιτύχουμε καλύτερο επιμερισμό των καθηκόντων. Αυτό προς επίρρωση των εφισταμένων διατάξεων ως προς το συντονισμό των δωρήτων για να αποφύγουμε τις περίτες και επικαλυπτόμενες διαδικασίες. Οποιαδήποτε δράση σε αυτό το τομέα θα πρέπει να παρακολουθείτε εκ του και να βασίζεται σε αποδείξεις, σε τεκμήρια. Ε, και άρα πρέπει ο κανονισμός να κωδικοποιεί τα μέτρα χάρη στα οποία θα μετρούμε την πρόοδο για τον αυξημένο συντονισμό των δωρητών και θα συμπεριλαμβάνουμε σχετικές πληροφορίες όπως παραδείγματο χάρη μια ομαδοποιημένες προφορίες για όλες τις ροές αναπτυξιακής βοήθειας, ε, διατάξεις σε σχέση με το εργατικό δίκαιο, ε, πρόθεση να μετάσχει κάνει τον σχεδιασμό των δράσεων, ε, δράσεις για να μειωθεί το κόστος των συναλλαγών και δέλτα, mainstreaming, του, των διαδικασιών στρατηγικού σχεδιασμού και επιμερισμού των καθηκόντων. Η διαφάνεια και ε, η δημοκρατική διαδικασία ανάπτυξη ενδογενών ικανοτήτων για αυτέ τι χώρε είναι απαραίτητα στοιχεία, ώστε να μετάσχουν όλο και περισσότερο τα εθνικά κοινοβούλια σε αυτή τη διαδικασία των διεθνών δωρητών. Ε, πρόεδρε, αν ένα πράγμα μπορούσαμε να κάνουμε θα ήταν να ενισχύσουμε τη συνεργασία ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια, ώστε να μπορέσουμε να επιτύχουμε το εξή. Τα Εθνικά Κοινοβούλια να έχουν τη δυνατότητα να επανέρχονται στα, ε, στις εν λόγω χώρες και να τις ενημερώνουν για τις ανασυχίες μας. Δεν είναι δική μας δουλειά ε, αυτή. Εκείνοι πρέπει να ε, αναλάβουν αυτή την ευθύνη. Και θα έπρεπε να δούμε να διαρευνήσουμε άλλους τρόπους συνεργασίας ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια. Ε, κοινέ αποστολέ και ε, πρέπει να γίνονται για να ε, αποτιμάται η πρόοδος και να συζητούμε τα πεπραγμένα και τα αποτελέσματα. Η αρχή της διαφάνειας και του δημοκρατικού ελέγχου ε, σημαίνει επίσης ότι θα συμμετέχουν και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα έξω και μία σύσταση στα πλαίσια του οργάνου, για την αναπτυξιακή βοήθεια, το DCI, καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μετρά την πρόοδο ε, που έχει σημειωθεί και τα μέτρα που έχουν υλοποιηθεί και να υποβάλει συνέχεια έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή των Περιφερειών αλλά και στην ΕΟ και Έχουμε και τη σύσταση υπαριθμών 9, όπου αναφέρεται μια ετήσια έκθεση για την υλοποίηση και όπου ε, προσμετρώνται τα αποτελέσματα τη αναπτυξιακή πολιτική. Δεν προσπαθούν, ε, δεν προσπαθεί κανεί να μα πάρει την εξουσία. Είναι συνδυασμένη η προσπάθεια όλων. Ε, ο καθένα κάτι διαφορετικό έχει να κάνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα καταθέτει προτάσει για τον συντονισμό. Ε, θα καταθέσει μάλλον προτάσει μέχρι το, την 31η Δεκεμβρίου του 2015 είναι λογικό το χρονοδιάγραμμα. Για θα έχει βγει και το νέο κοινοβούλιο. Τι θα γίνει τώρα το επερχόμενο κοινοβούλιο θα πρέπει να μπορεί να επεξεργαστεί μία πρόταση που θα έχει καταθέσει λίγο νωρίτερα, όχι πολύ νωρίτερα, λίγο νωρίτερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ούτω ώστε να ληφθούν δεόντω υπόψη οι απόψει τη Επιτροπή Ανάπτυξη και τη Ολομέλεια. Σαν κατακλείδη, Πρόεδρε, αυτή η πρωτοβουλία δεν πρέπει να θεωρηθεί ω ένα πρόσκομα σε σχέση με τι μέχρι τούδε προσπάθειε ε, του ε, Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξη και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα πρέπει να ε, κληθούν ω θετικέ και να υποστηριχθούν από όλου. Το αντίθετο χρησιμοποιούμε ε, πολιτική μόχλευση αν ακολουθήσουμε αυτές τις προτάσεις για να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα ούτω ώστε να γίνονται σεβαστέ και οι δεσμεύσει για την αναπτυξιακή βοήθεια και η χορήγηση αναπτυξιακή βοήθεια. Λοιπόν, η χρηματοπιστωτική μόχλευση τη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, δράζεται επί των μεμονωμένων δράσεων των 28 κρατών μελών καθώ και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Euh, Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μίτσελ, για αυτή την παρουσίαση τη έκθεσή σα. Γνωρίζουμε όλοι ότι προφανώ τα κονδύλια θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν πολύ καλύτερα ιδιαίτερα, ιδιαίτερα σε μια εποχή κρίση που βιώνουμε αυτή τη στιγμή. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα δώσω τώρα το λόγο στους βουλευτέ που τον ζήτησαν, Κεραίρο Σαλόμο. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ θα ήθελα απλά να μου επιτρέψετε να σχολιάσω λίγο θετικά την έκθεση την οποία μας παρουσιάζεται λόγω ακριβώς της πεποίθησης την οποία έχετε και, και τη στάση που επιδείξατε επίσης και στις διμερείς επαφές που απέδειξαν ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε σε αρκετά θέματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα αυτό γιατί στα πλαίσια της συγκυρίας συμπίπτουν δύο κομβικά θα έλεγα σημεία. καταρχά η μείωση της βοήθειας για την ανάπτυξη, μείωση της δημοσιονομικής βοήθειας δηλαδή από διάφορες χώρες. Κάποιες από τις χώρες αυτές έχουν σοβαρά προβλήματα στα δικά τους οικονομικά και υψηλά ελλείμματα. Και άλλες χώρες απλά εποφελούνται από την κατάσταση για να μειώσουν τη συμμετοχή τους και την εμπλοκή τους στην ανάπτυξη και συνεργασία. Έχουμε πάντως ε, μία φάση μειωμένων εσόδων και δεν θα κλείσει η φάση αυτή αρκετά γρήγορα, από ό,τι φαίνεται θα παραταθεί ε, επί Ταυτόχρονα υπάρχει μία ανάλυση η οποία έχει γίνει σχετικά με τη διασπορά των προσπαθειών μας. Ανάλογα με τους τομείς θεματική δηλαδή διασπορά, χωρική διασπορά, που τελικά μειώνει το βάρος της παρέμβασής μας και την προσπάθεια επίτευξης των στόχων που επιδιώκουμε και που κυρίως ε, είναι η μείωση της ένδυας. Τα στοιχεία τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας και τα οποία προέρχονται από διαφορετικού τύπου μελέτες δεν συμπίπτουν όλα βέβαια μεταξύ τους, αλλά τίνουν σίγουρα προς την ίδια κατεύθυνση. Η κατεύθυνση αυτή λέει ότι η διασπορά και η έλλειψη συντονισμού μειώνει ουσιαστικά τη δυνατότητα παρέμβασής μας επί της ουσίας. Δεν υποστηρίζω εγώ ούτε και η ομάδα μου ότι θα πρέπει να κάνουμε περισσότερα με λιγότερα, γιατί δεν θέλουμε να έχουμε λιγότερα. Το θέμα είναι να επιδιώξουμε περισσότερα αλλά με τα ίδια οικονομικά τουλάχιστον μέσα. Αυτή θα πρέπει να είναι η προσπάθεια, να αυξήσουμε δηλαδή τα αποτελέσματα με τα ίδια ποσά στη διάθεσή μας. Αυτό μπορούμε να το πετύχουμε και με μια καλύτερη συνεργασία και θα ήθελα να μάθω ακριβώς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας κάνει προτάσεις για διάφορους μηχανισμούς έτσι ώστε να μπορέσουμε να αυξήσουμε το επίπεδο συνεργασίας μας, έτσι ώστε η συνεργασία μας αυτή να μην εξαρτάται αποκλειστικά από την βούληση του καθενός από τα κράτη-μέλη, αλλά να υπάρχουν στοιχεία, θα έλεγα, αναγκαστικού χαρακτήρα υποχρεωτικότητας που να λειτουργούν σαν κίνητρα έτσι ώστε να υπάρξει μια τέτοια μορφή καλύτερου συντονισμού. Το πρόβλημα το οποίο συναντάμε εδώ δεν είναι ένα νέο πρόβλημα, το γνωρίζουν όλοι. Πάρα πολλές από τις χώρες μας έχουν διαφορετικού τύπου συμφέροντα. Μερικές φορές οι ίδιες αυτές οι χώρες κάποιες περιοχές του κόσμου τις θεωρούν ιδιαίτερο συγγενείς και γι' αυτό ακριβώς τις προωθούν κατά προτεραιότητα. Άλλοι πιστεύουν ότι έχουν, ε, ε, θα έλεγα, μια ειδική ευαισθησία απέναντι σε κάποιες χώρες τις οποίες θα ήθελαν να αναπτυχθούν και αυτό δημιουργεί κάποιους εγωισμούς στη συμπεριφορά των κρατών μελών που επηρεάζουν αρνητικά τα αποτελέσματα τα οποία πετυχαίνουμε. Συνειδητοποιούμε πάντως ότι εμείς δεν είμαστε σε θέση να διαγράψουμε πλήρως την επιθυμία, την πρόκληση των κρατών μελών να καλύψουν ένα συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο, επί τη βάση της ευαισθησίας ή των ειδικών χαρακτηριστικών. Απλά πρέπει αυτή την ευαισθησία, αυτή την πρόκληση να την εντάξουμε στους μηχανισμούς συντονισμού. Στα πλαίσια της μελέτης που έγινε από τρία think tank, τα οποία γνωρίζουμε, μας δίδει ορισμένα στοιχεία και περιλαμβάνει και ορισμένες προτάσεις για την εντατικοποίηση του συντονισμού σε διάφορα επίπεδα, να ενισχυθούν οι βέλτιστες πρακτικές, να εκμεταλλευτούμε τις δυνατότητες συντονισμού ακριβώς σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους χαρηγείται η βοήθεια και να μπορέσουμε να βοηθήσουμε καλύτερη χωρική κατανομή των ε, ε, προϊόντων, αν θέλετε, της προσπάθειας την οποία κάνουμε μέσω του καλύτερου συντονισμού. Ο δρόμος τον οποίο χαράζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι σαφής, είναι καλύτερη μορφή συντονισμού. Βασικός στόχος είναι, είναι αν θέλετε εκεί που θέλουμε όλοι να φτάσουν, είναι το λιμάνι στο οποίο θέλουμε όλοι να καταλήξουμε, δηλαδή κοινοτικοποίηση της αναπτυξιακής βοήθειας. Είναι προφανές ότι μπορεί να υπάρχουν διαφορές μέσα από τις φάσεις και τα στάδια τα οποία πρέπει να περάσει κανείς για να καταλήξει σε αυτό τον τελικό στόχο και γι' αυτό ακριβώς είναι απαραίτητο να ακολουθήσουμε έναν στρατηγικό χάρτη, ένα οδικό χάρτη, έτσι ώστε μέσω των αυξανόμενων προσπαθειών στα διάφορα επίπεδα συντονισμού να τίνουμε όλοι επιμένω προς την ίδια κατεύθυνση και προς ένα τελικό αποτέλεσμα που είναι ακριβώς η κοινοτικοποίηση της αναπτυξιακής συνεργασίας. Εγώ εξήγησα στον κύριο Μίτσελ ότι η πολιτική μου ομάδα δεν είναι καθόλου κατά σε κάποια φάση να καταλήξουμε ακριβώς στο να είναι υποχρεωτικό νομικά θα έλεγα να υπάρξει ένα ρυθμιστικό μέσο Instrument y que eh, tenemos todavía que είναι κάτι το οποίο είμαστε διατεθαμένοι να συζητήσουμε, να αντιμετωπίσουμε. Αυτό δεν ξέρω αν θα το επιδιώξουμε τώρα ή θα είναι ακριβώς αποτέλεσμα ενός οδικού χάρτη τον οποίο θα πρέπει να ακολουθήσουμε πάντως, όπως ακριβώς έχει ήδη υπογραμμίσει ο κύριος Μίτσελ, το 2015 θα έλεγα είναι ένα χρονικό πλαίσιο επαρκές έτσι ώστε να παρουσιάσει τις προτάσεις της Ευρωπαϊκή Επιτροπή όχι μόνο γιατί θα έχει υπάρξει ένα νέο εκλεγέν κοινοβούλιο αλλά και μια νέα επιτροπή. Και έτσι θα έχει ελπίζουμε αλλάξει προς το καλύτερο και η οικονομική κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί ε, ίσως ε, σε αυτή την περίπτωση να υπάρχει και ανάκαμψη της αναπτυξιακής βοήθειας σε οικονομικούς όρους. Ευχαριστώ λοιπόν τον κύριο Μίτσελ για την έκθεσή του. Νομίζω ότι επί της ουσίας συμφωνούμε πλήρως μαζί σας. Και συμφωνούμε επίσης στην προσπάθεια να βρούμε ένα κοινό δρόμο για να πετύχουμε αυτό το στόχο. Ευχαριστώ πολύ. Η Ρενάτε Χάλεν της Γενικής Διεθνής Λεύκο έχει το λόγο. Good afternoon, many thanks. Καλό απόγευμα, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πρώτα πρώτα για το ενδιαφέρον που επιδεικνύει το Κοινοβούλιο να βελτιώσει το συντονισμό και πραγματικά αυτός είναι και δικός μας στόχος στον οποίο έχουμε επενδύσει εδώ και πολλά χρόνια. Εσείς αναφέρεστε εδώ σε πάρα πολλά έγγραφα αναφοράς τα οποία υπάρχουν και αυτό ακριβώς δείχνει πόσα χρόνια ασχολούμεθα με, το θέμα για να βελτιώσουμε με την υπόθεση αυτή για να βελτιώσουμε τον συντονισμό έχουμε μια ε, ενωσιακή πολιτική ανάπτυξη που είναι παράλληλη με τη, αυτή των κρατών μελών αλλά βεβαίως σε πολλά κράτη-μέλη υπερισχύουν τα εθνικά συμφέροντα. Συμφωνώ με την ιδέα να ευρωπαϊκοποιήσουμε κατά κάποιο τρόπο την ευρωπαϊκή βοήθεια αλλά πιστεύω ότι επουδενή λόγο μπορούμε να φιλοδοξούμε ότι θα επιτύχουμε ε, κοινοτική ε, πολιτική. Αυτό δεν συμβαδίζει και με τη συνθήκη. Αλλά γενικώ να ενισχύσουμε την ένωση, να ενισχύσουμε, να βοηθήσουμε τις χώρες όταν δρούμε, ε, αναλαμβάνουμε δράση επί του πεδίου. Αυτό σίγουρα. Στα προπαρασκευαστικά έγγραφα λέγεται και το τονίζω ότι μας ανησυχεί ένα πράγμα αν κωδικοποιήσουμε νωρίς ε, το να κωδικοποιήσουμε πολύ ο, το, από τώρα τη το πώς θα προχωρήσει το πρόγραμμα, το να ευθυγραμμίσουμε αυτά που θέλουμε να κάνουμε μαζί με τις χώρες μέλη, να ε, παρακολουθούμε πραγματικά εκ παραλλήλου τη δουλειά που γίνεται αυτό πραγματικά είναι κάτι το είναι ένα μεγάλο άλμα το οποίο πρέπει να γίνει ήδη έχουμε κάνει αρκετές πρόοδους θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε ε, και ε, είμαστε σίγουροι ότι θα επιτύχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Εσείς τώρα μιλάτε για ένα νομοθέτημα δεσμευτικό από νομικής απόψεως. Προτρέχετε τρόπον την να... Ε, δεν ξέρω αν αυτό είναι καλό γιατί και η δική μας ε, διαδικασία αποδίδει καρπούς και προχωρούμε παράλληλα όπως είπα. Δεν μπορούμε να πιέσουμε παραπάνω τα κράτη-μέλη. Εκείνο όμως το οποίο θα ήταν καλύτερο από αυτό που προτείνετε εσείς για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τα κοινά προγράμματα που ξεκινούν και το, τον οποίο ο αριθμός θα αυξηθεί τις επόμενες χρονιές εκείνο λοιπόν που μπορούμε να κάνουμε και για το οποίο πραγματικά θα σας είμαστε ευγνώμονες και που θα ήταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έρθει σε μεγαλύτερη σύνδεση σε στενότερη σχέση με τα εθνικά ε, κοινοβούλια και τις εθνικές αρχές για να ρωτήσει για να ε, κανονίσει τι θα μπορούσε να γίνει για να μπορέσουν και περισσότεροι να συνεργαστούν για να μπορούμε να μιλούμε όλοι με μια φωνή. Αυτό θα μπορούσε να γίνει εδώ, να μπορούσε να γίνει στα εθνικά κοινοβούλια και όπως σας είπα υπάρχει ήδη κάποια πρόοδος αλλά είναι γεγονός ότι ε, βλέπουμε όλο και περισσότερο ότι χρειάζεται να καλούμε ε, τους προϊσταμένους μας να συζητούμε την πρόοδο και τα επιτεύγματα τους χάνει, στα κοινά προγράμματα. Αν διαβάσετε τη συνθήκη το 2010 άρθρο δεν αναφέρεται μοναχά στο συντονισμό μέσω των κοινών προγραμμάτων. Πάει λίγο παραπέρα η συνθήκη. Μιλάει για το συντονισμό τομέων στο εσωτερικών χωρών. Και βλέπουμε τώρα τα κράτη-μέλη όντως να ενδιαφέρονται να γίνει κάτι τέτοιο. Και πιστεύουμε ότι γίνεται με αυτόν τον τρόπο και καλύτερη κατανομή εργασίας στις διάφορες χώρες αλλά πρόκειται για μια διαδικασία που ακολουθεί το ρυθμό της δεν είναι ταχεία διαδικασία αλλά προχωρεί και κάτι τι άλλο υπάρχει που πραγματικά είναι έρχεται φυσικά και δεν απαιτεί τίποτα να κάνει η Κομισιόν. Ε, όταν ετοιμάζουμε τις θέσεις μας για τις, για τις διεθνείς συσκέψεις εκεί που δεν ξέρουμε καν που δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει ενιαία θέση από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης εκεί λοιπόν ε, βλέπουμε ότι παρόλο που είναι προαιρετικό οι θέσεις είναι πολύ παρόμοιες και θα μπορούσαν να είναι ενιαία η θέση θα ήθελα να σταματήσω εδώ, δεν χρειάζεται να πω τίποτα παραπάνω. Ξέρω ότι ο συνάδελφος από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ε, πάρει το λόγο. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Δίνω το λόγο στον κύριο Αλέξη Ζεμπραντή. Λέγομαι Άλεξ Χεμπράντη και είμαι Ολλανδός. Σας ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο. Να ευχαριστήσω και την, Ευρωπαϊκή, την Επιτροπή σας για την προσπάθεια την οποία κάνατε και κυρίως τον κύριο Μίτσελ. Θα ήθελα να υπογραμμίσω τη στενή συνεργασία που έχουμε με την ΤΕΦΚΟ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα ήθελα να βασίσω τα σχόλιά μου και στα δικά τους. Τέσσερα σημεία. Καταρχάς υποστηρίζουμε την ανάλυση και τα συμπεράσματα της έκθεσης ότι δηλαδή απαιτείται ενισχυμένη συνεργασία η οποία ε, σαν προσπάθεια την έχουμε ξεκινήσει ήδη από το 1974 ε, και προσπαθούμε να προχωρήσουμε. Και υπάρχει φυσικά και πολύ σημαντικός ρόλος και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για τα κράτη-μέλη έτσι ώστε ε, να ελέγχονται σωστά οι συμπεριφορές από πλευρά των κρατών μελών. Σεβόμαθε πλήρως ε, την ηγετική θέση την οποία έχει βέβαια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με τον προγραμματισμό και τον αποκοινού προγραμματισμό. Και αυτό το οποίο θα θέλαμε να προτείνουμε είναι να υπάρξει, θα έλεγα, μια, να χρησιμοποιήσουμε την απόφαση του Ιουλίου του 2010, όπου αποφασίζεται και η δημιουργία της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης. Θα θέλαμε επίσης να υπογραμμίσουμε το θέμα του κοινού προγραμματισμού, και θα θέλαμε αυτό να αντικατορπίζεται καλύτερα στην έκθεση και αυτό για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί πιστεύουμε ότι ο κοινό προγραμματισμός έχει ήδη παρουσιαστεί σαν ε, το θέμα με το μεγαλύτερο δυναμικό, αν θέλετε, για τη βελτίωση της ε, αποδοτικότητας, ε, προστατεύει γενικά τις αρχικές πρωτοβουλίες μονομένων χωρών, αλλά συντονίζει κιόλας, αυξάνει τον έλεγχο γενικότερα και όπως είπε και ο συνάδελφος από την ΤΕΦΚΟ θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η διαδικασία αυτή προσφέρει πολύ περισσότερα από ό,τι στο παρελθόν. Έχουμε άνω των 40 χωρών μέσω κοινών προγραμμάτων για τις μισές αυτές ξεκινάμε ήδη είτε φέτος είτε του χρόνου, σύντομα δηλαδή. Έχουμε ήδη τα πρώτα αποτελέσματα από Γουατεμάλα, το Λάος, την Ουγκάντα και άλλες περιπτώσεις και έχουμε επίσης ε, και περιφερειακά τέτοια προγράμματα συντονισμού, όχι μόνο για χώρες ε, χαμηλού εισοδήματος, αλλά και για τις λεγόμενες εύθραυστες χώρες. Νομίζω ότι μπορούμε να καλύψουμε με τον τρόπο αυτό το 70 περίπου της 100 μέσω του κοινού προγραμματισμού δηλαδή. Προτείνουμε επίσης να υπάρξουν κάποιες αναφορές στον κοινό προγραμματισμό, στο έγγραφο το οποίο προτείνει ο κύριος Μίτσελ. Το τελευταίο θέμα που θέλω να θέσω αφορά το χρονοδιάγραμμα το οποίο έθεσε και η συνάδελφος της ΔΕΦΚΟ. Ίσως εδώ να απαιτείται κάπως περισσότερη συζήτηση. Ο κοινός προγραμματισμός ξεκίνησε θα έλεγα ε, ε, τώρα ουσιαστικά και είναι ένα μέσο ευέλικτο για τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίζουμε τα θέματα των διαφόρων χωρών. Έχουν γίνει κάποια βήματα τον τελευταίο χρόνο εγώ είμαι για 10 χρόνια εδώ σε αυτή την υπηρεσία και για πρώτη φορά βλέπω ότι έχουν υπάρξει βήματα πρόοδου. Γιατί πέρα από την προσπάθεια την οποία κάνουμε έτσι και αλλιώς σε ε, πολιτικό και σε λειτουργικό επίπεδο έχουν υπάρξει σημαντικά βήματα προόδου. Η συνθήκη της Λισαβόνας βοηθά στη συνεργασία και στην προσφυγή στον κοινό προγραμματισμό. Δεν πρέπει επίσης να υποτιμάμε και το ρόλο των αντιπροσωπιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος είναι κομβικός, είδαμε ότι ήδη έχουν κάνει πάρα πολλά και έχουμε επενδύσει και αρκετά στην προσπάθεια γεφύρωσης των διαφορών ανάμεσα στις αρχικές δεσμεύσεις ε, ε, πιστώσεων και στις τελικές πιστέσεις οι οποίες χρησιμοποιούνται. Τέλος υπάρχουν και ε, ε, θα έλεγα εξωτερικοί παράγοντες οι οποίοι και αυτοί μας πιέζουν ε, στο να προχωρήσουμε σε καλύτερες μορφές συντονισμού. Προσπαθούμε λοιπόν να συνεργαστούμε όσο καλύτερα μπορούμε και με τις καινούργιες ισχυρά οικονομικές χώρες, αναδυόμενες οικονομίες που και αυτές συμμετέχουν θα πρέπει λοιπόν να θεωρήσουμε λίγο το χρονοδιάγραμμα, να μας δώσετε την δυνατότητα να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο στα πλαίσια του κοινού προγραμματισμού και να βγάλουμε τα κατάλληλα συμπεράσματα. Σας ευχαριστώ για μια ακόμη φορά για την δυνατότητα που μας δώσατε να είμαστε παρόντες εδώ. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Κουάκενμπος ε, του δικτύου Concord, έχετε το λόγο. Hello. Um, Ευχαριστώ. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσω ενώπιόν σας και θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Ε, Γενικότερα μιλώντας, θα συμφωνήσουμε τόσο με την ε, φρασιολογία, τη διατύπωση, όσο και το περιεχόμενο της έκθεσής μας αρέσει η έμφαση που δίνει στο σύστημα των κρατών μελών, την ευθυγράμμιση των εθνικών στρατηγικών. Είναι άριστη η ιδέα και καλύπτει πολλές ανησυχίες που έχουμε για τον συντονισμό, ε, για το, την επίτευξη ισορροπίας ανάμεσα στις χώρες δωρητές και στις χώρες δικαιούχους. Θα θέλαμε επίσης ε, βεβαίως να τονίσουμε τους περιορισμούς για όλους, όχι μόνο για τα κράτη-μέλη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ε, θα έχει για τα επόμενα χρόνια χρηματοδοτήσει οικονομικούς περιορισμούς και τι σημαίνει αυτό για την υλοποίηση του κανονισμού και ποιοι πόροι θα είναι διαθέσιμοι για τη χρηματοδότηση της δράσης που προτείνει. Το μήνυμά μας είναι μια ξεκάθαρη αναφορά στην αρχή της, του democratic ownership, της ε, ανάπτυξης των ικανοτήτων των ίδιων των χωρών Επίσης θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι η συνοχή και η αποτελεσματικότητα ε, θα πρέπει να επιδιώκονται για την αναπτυξιακή βοήθεια και αυτό να μην σχετίζεται με τις ε, στρατηγικές προτεραιότητες οι οποίες θα πρέπει να αποφασίζονται από την ίδια τη χώρα δικαιούχο. Σας ευχαριστούμε. Θα ξανακούσουμε και πάλι τον κύριο Μίτσελ ε, για τις καταληκτικές παρατηρήσεις. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον ε, συνάδελφο Γκερέρο ε, για τα επικοδομητικά του σχόλια και την υποστήριξη που μου προσφέρει για το βασικό περιεχόμενο της έκθεσης. Φυσικά θα πρέπει να προσαρμόσουμε κάποιες λεπτομέρειες, αλλά έχουμε άπλητο χρόνο για τις ε, τροπολογίε ε, και συνενετικές λύσεις και σίγουρα θα καταλήξουμε σε αυτές. Πάντως συμφωνούμε για τη γενική προσέγγιση και αυτό είναι θετικό. Σε σχέση τώρα με τα σχόλια τη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ ΝΤΕΦΚΟ και τη υπηρεσία εξωτερική δράση, η επίτευξη τη σωστή ισορροπία. Όντω, αυτό χρειαζόμαστε Όμω, ε, όμως, ε, τίθεται το ερώτημα, είναι η σωστή στιγμή εμείς δεν προτείνουμε να έχουμε δεσμευτική αναπτυξιακή βοήθεια. Μπορούμε να έχουμε μια νομοθετική πρόταση ε, που να ε, ε, χαρακτηρίζεται από ήθος, από την αρχή της συνεργασίας κτλ. Ωραία. Και σίγουρα κάποια στοιχεία πρέπει να είναι δεσμευτικά, αλλιώς δεν πρόκειται κανείς να κάνει τίποτα. Αλλά το θέμα είναι ο χρονισμός. Μιλάμε για το 2015. Τι θα κάνουμε. Αν χάσουμε και αυτό το πλοίο θα πάμε για τις επόμενες εκλογές Ε, πάντως νομίζω ότι ε, μπορούμε να επιτύχουμε την ισορροπία που θέλουμε και στο άρθρο 310 της συνθήκης λέει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να αναλάβει αδίποτε ε, πρόσφορη πρωτοβουλία για να συντονίσει τη δράση των κρατών μελών στον τομέα της αναπτυξιακής πολιτικής. Οπότε το βασικό μας επιχείρημα είναι ακριβώς αυτό. Έχουμε βάση, νομική βάση για την έκθεση. Και ως προς τον κοινό σχεδιασμό ανοιχτοί είμαστε. Αυτό που μας πρότεινε εξωτερική δράση, η υπηρεσία εξωτερική δράσης, μπορείτε να μας στείλετε τα σχόλιά σας και να τα εξετάσουμε. Ε, σε σχέση με τον, αυτά που είπε ο εκπρόσωπος ε, του Concord, ε, ε, χαίρομαι με τα σχόλια για τη διατύπωση και θα συμφωνήσω ότι χρειάζεται και η διαφάνεια και αυτό το democratic ownership και σίγουρα πρέπει να συνεργαστούν όλα τα θεσμικά όργανα, αλλά ξέρετε η Επιτροπή των Περιφερειών και η ΕΟΚΕ Καθώς και η Επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 9 για την υποβολή σε έκθεση, καλά αυτό θα το δούμε στο πεδίο εφαρμογής, και ούτως ή άλλως θα δούμε ποιες ελλείψεις έχει διατύπωση, αλλά ξαναλέω ότι η διαφάνεια και το democratic ownership είναι ε, απαραίτητα στοιχεία. Ε, σίγουρα πιστεύουν όλοι ότι χρειάζεται καλύτερο συντονισμός. Τώρα ας δούμε και το χρονοδιάγραμμα. Ελπίζω να είναι βαθιές οι ρίζες της οικονομικής ανάκαμψης και άρα ε, θα έχουμε τους απαιτούμενους πόρους για να προχωρήσουμε. Το πώς θα τους χρησιμοποιήσουμε τους πόρους είναι αυτό που έχει σημασία για να καλυφθούν οι καθημερινές ανάγκες ε, των ε, πλέον απόρων αυτού του πλανήτη. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να καταλήξουμε σε μια συνενετική λύση και ας ελπίσουμε ότι θα είναι καλή η έκθεση. Αλλά πάντως αυτή η ομοθυμία εδώ στο Κοινοβούλιο μπορεί να εξυπηρετήσει έναν ευγενή στόχο. Θα ήθελα να ευχαριστώ όλους όσους με βοήθησαν ε, για να συντάξω την έκθεσή μου. Σας ευχαριστούμε για την κατάθεση τροπολογιών για το σχέδιο έκθεσης. Έχουμε τη 10η Οκτωβρίου ως καταληκτική ημερομηνία μέχρι τις 12 και στις 5 Νοεμβρίου θα γίνει ψηφοφορία. Τώρα θα κάνουμε μια συντομότατη διακοπή γιατί είμαστε πολύ γρήγοροι. 5-10 λεπτάκια για να υποδεχτούμε τον επίτροπό μα. Δεν έρχονται και κάθε μέρα. Voilà. Donc nous attendons... Περιμένουμε τον Επίτροπο Πίμπαλξ και τον κύριο Ποτόσνικ, ε, Επιτρόπους για θέματα ανάπτυξης και για θέματα περιβάλλοντος και την κυρία Αμίνα Τζέι Μοχάμε, τη δική σύμβουλο του Γενικού Γραμματέα του ΕΕ σχετικά με τον προγραμματισμό της ανάπτυξης του 2015, 5-10 λεπτά για διακοπή και συνεχίζουμε.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 Alors, mes chers collègues, nous abordons... Λοιπόν, ε, συνάδελφοι, φτάνουμε σε ένα κομβικό θέμα για την ανάπτυξη μέσα σε ένα υγιές περιβάλλον και θα προσπαθήσουμε να δώσουμε απαντήσεις ε, και για τη δική μας Επιτροπή αλλά και για άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές που συμμετέχουν για τους στόχους της αηφόρου ε, ανάπτυξης και για τους στόχους της χιλιετίας για την ανάπτυξη με τους επιτρόπους Πίμπαλξ και Ποτότσνικ που είναι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη και το περιβάλλον. Τους καλωσορίζω με χαρά σήμερα. Θέλουμε να συζητήσουμε πριν από την 68η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον που θα οργανωθεί στις 25 Οκτωβρίου, Σεπτεμβρίου συγγνώμη, έτσι ώστε να συμπέσουν οι στόχοι για την αηφορία με τους στόχους για τη χιλιετία. Ε, θα ήθελα επίσης να καλωσορίσω τους δύο, να καλωσορίσω και την κυρία Αμινά Μοχάμεντ, ειδικό σύμβουλο του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών υπεύθυνη για το πρόγραμμα που καταλήγει το 2015 που με μεγάλη χαρά την καλωσορίζουμε σήμερα για μια ακόμη φορά. Ευχαριστώ επίσης και τους συναδέλφους της Επιτροπής Περιβάλλοντος και κυρίως τον πρόεδρό της, τον κύριο Ματίας Γκρότε. Θα ήθελα να ξεκινήσω δίδοντας το λόγο στον συνάδελφο ε, πρόεδρο της Επιτροπής, ε, τον κύριο Γκρότε. Και μετά θα πάρουν το λόγο οι δύο επίτροποι. Κύριε συνάδελφε, σας ακούμε. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, συνάδελφοι, εξαιότιμη κυρία Μοχάμεντ, κύριοι Επίτροποι, ειδικά τον κύριο Ποτότσνικ τον συγχαίρω για το βραβείο. Χαιρόμαστε που ε, δικαίως πήρε το βραβείο αυτό. Στην ε, ημερήσια διάταξη έχουμε τα θέματα που αναφέρατε κυρία Πρόεδρε και τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά ε, και είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε την συνεδρίαση αυτή που κάνουμε αν θέλουμε να εφαρμοστούν κάποια στιγμή οι αναπτυξιακοί στόχοι της χιλιετίας. Θα πρέπει να συζητήσουμε ε, ορισμένα πράγματα. Προ, ε, προετοιμάζοντα το Ρίο Συνήκωση ε, συζητήσαμε συναφή θέματα. Ο κύριος Νόιτσερ ε, με τον κύριο Νόιζερ συζητήσαμε πολύ. Ε, έβγαλε και ένα βιβλίο ο κύριος Νόιζερ σχετικά με το πώς θα μπορούσαμε να εφαρμόσουμε τους στόχους αυτούς της ε, χιλιετίας γιατί πολλές φορές μας κατηγορούν ότι δεν προχωρούμε αρκετά γρήγορα ε, τελικά το θέμα δεν είναι αν ακολουθούμε εμείς τον υπόλοιπο κόσμο όσον αφορά το, ρυθμό μας ή το αντίθετο. Εκείνο που είναι σημαντικό είναι να προετοιμαζόμαστε καλά και με πράσινη υπο, πράσινες υποδομές, με ανανεώσιμες ενέργειες και με ε, ε ενθουσιασμό να εφαρμόσουμε, να κάνουμε ορισμένα πράγματα στον πλανήτη μας ούτω ώστε μετά το 2015 να έχουμε αυτά αποτελέσματα. Γι' αυτό θεωρώ ότι η σημερινή συζήτηση είναι πολύ σημαντική. Τώρα η συνδιάσκεψη Ρίο συνήκωση ε, απέδωσε περισσότερους καρπούς από ό,τι περιμέναμε αλλά λιγότερους από ό,τι ελπίζαμε. Έτσι θα περιέγραφα τα αποτελέσματα του συνδιάσκεψης αυτής. Ε, περιπτώσει χαίρομαι που θα γίνει η συζήτηση ε, σας ευχαριστώ που ήρθατε όλοι πιστεύω ότι πρέπει να ανασκουμποθούμε όλοι γιατί είναι Ηράκλειος ο άθλος που μας περιμένει και η δική μας επιτροπή έχει ακόμη πιο πολλά πράγματα να κάνει από τι άλλες επιτροπές Ευχαριστώ. Δίνω το λόγο στον κύριο Πίμπαλξ, στον Επιτρόπο για 8 λεπτά. είναι ιδιαίτερα επίκαιρο το ζήτημα και πάρα πολύ σημαντικό να γίνεται μεικτή συνεδρίαση των δύο επιτροπών. Θα αναθεωρηθούν οι στόχοι της χιλιετίας από τον ΟΗΕ και θα συζητηθεί το επόμενο πλαίσιο τώρα. Ε, οπότε είναι ιδιαίτερα επίκαιρη η μεικτή συνεδρίαση. Επίσης αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του ότι, ε, της δέσμευσης μάλλον που έχει αναλυθεί για την ε, οικοδόμηση ενός θεματολογίου για την περίοδο μετά το 2015 για την εκρίζωση της ε, φτώχειας και για την διασφάλιση της αηφόρου ανάπτυξης στον πλανήτη μας. μετά το 2015 επιδιώκεται ένα συνολικό πλαίσιο, ποτέ θα εκκριζωθεί η φτώχεια εάν δεν ακολουθήσει μια βιώσιμη πορεία ε, ο πλανήτης Γη με τρόπο ώστε να αντιμετωπίσουμε τις κλιματικές ε, αλλαγές. Ε, αυτό είναι ένα θέμα που ενδιαφέρει όλους τους πολίτες. Είναι πάρα πολύ σημαντική η συμβολή σας, η έκθεση Κατσμάρεκ, το ψήφισμα που ενέκρινε τον Ιούνιο ε, το Κοινοβούλιο για τους στόχους της χιλιετίας και του προσδιορισμού του πλαισίου μετά το 2015. Ε, αυτά ενίσχυσαν σε σημαντικό βαθμό την θέση και το ειδικό βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διεθνή σκηνή. Ας κοιτάξουμε τώρα πώς διαμορφώνει το γενικό πλαίσιο του 2015. Για να προσδιοριστεί αυτό το πλαίσιο πρέπει να αντιμετωπίσουμε δύο βασικές προκλήσεις για να επιτύχουμε ό,τι είναι επιτεύξιμο και το γνωρίζουμε όλοι. Μια καλύτερη ζωή για όλους. Αυτή η ειδική εκδήλωση για τους στόχους χιλιετίας θα ευαισθητοποιήσει την διεθνή κοινότητα ούτω ώστε να καταλήξει σε συμφωνία για το θεματολόγιο μετά το 2015. Κατά τη γνώμη μου η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ζητήσει παγκόσμια δράση σε δύο μέτωπα. Πρώτον, πρέπει να ολοκληρώσουμε αυτά που αρχίσαμε, δηλαδή στις προσπάθειες που κάνουμε για την επίτευξη των στόχων της χιλιετίας ε, δεν πρέπει να εγκαταλείψουμε τις προσπάθειές μας τα επόμενα δύο χρόνια. Η έκθεση του Γενικού Γραμματέου Μπάν και μου ζητά αξιοπρεπή διαβίωση για όλους και αναφέρει σημαντική πρόοδο για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας με υπερηφάνεια. Μπορώ να σας πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης έχει κάνει πάρα πολύ σημαντική συμβολή σε αυτή την πρόοδο για να μην πω τη σημαντικότερη. Τα τελευταία δέκα χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη τη ε, δέσμευσαν 50 δις το χρόνο για την αναπτυξιακή βοήθεια, άνω του ίμιση τη παγκοσμίου αναπτυξιακής βοήθειας. Ε, σας έχω ε, φέρει κάποια σχέδια του επικαιροποιημένου εγχειριδίου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής που θα δημοσιευθεί επίσημα την επόμενη εβδομάδα, όπου αναφέρεται λεπτομερώς για όλου τους στόχους της χιλιετία της Συμβολή Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό σημείο αναφορά και για τις δικές σας ε, εργασίες. Μέσω του EDF ε, ε, έχουμε εξασφαλίσει πρόσβαση σε πόσιμο νερό για 70 εκατομμύρια νοικοκυριά, 40 εκατομμύρια παιδιών έχουν πάει στο σχολείο, έχουν εμβολιαστεί, 20 εκατομμύρια παιδιά για μαγουλάδες, ευλογία και η Λαρά μάλλον και βλέπουμε ε, έμπρακτα την συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ταυτόχρονα παρακολουθείτε βήμα-βήμα τη δράση που αναλαμβάνουμε μέσα από αυτά ε, τα δύο όργανα όμως ε, υπερβολικά πολλές ε, γυναίκες ε, παλεύουν για να επιβιώσουν τον τοκετό, το ίδιο παλεύουν και τα παιδιά. Τα φάρμακα είναι πολυτέλεια για πολλούς, μπορούμε να κάνουμε περισσότερο. Ο Γενικός Γραμματέας Μπαν Κιμούν ρητά αναγνώρισε τον ηγετικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκρίζωση της φτώχειας στην πρόσφατη έκθεση που κατέθεσε εν ώψη αυτής της ειδικής εκδήλωσης. Θα επιδιώξουμε λοιπόν την υλοποίηση αυτών των στόχων ε, η πρωτοβουλία του Πρόεδρου Μπαρόσο για το 1 δίσε που ξεκίνησε το 2010 είναι ένα από τα βασικά εργαλεία που θα χρησιμοποιήσουμε για να επιτύχουμε τους στόχους μας. Για το προτινόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και η χρηματοδότηση που εξασφαλίζει για την αδειξιακή βοήθεια τελικά εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να αναδειχθεί στον πλέον γενναιόδωρο δωρητή και να συνεχίσει να διαδραματίζει αυτόν τον ηγετικό ρόλο ε, για την επίτευξη και των στόχων τη χιλιετία, αλλά και για τον προσδιορισμό του πλαισίου για την περίοδο μετά το 2015. Πάω στο δεύτερο μέτωπο τώρα. Θέλουμε ένα φιλόδοξο πλαίσιο για την περίοδο μετά το 2015. Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε μια αξιοπρεπής διαβίωση για όλου, θέτει ένα όραμα πόσο μπορούμε να συνδυάσουμε την εκρίζωση, την καταπολέμηση τη στόχη με την βιώσιμη ανάπτυξη. Υπάρχουν πέντε σημεία κλειδιά που έχουμε συζητήσει και σε προηγούμενη συνεδρίαση. Πιο συγκεκριμένα η ανάγκη για βασικές συνθήκες διαβίωσης έχουν τη δυνατότητα οι άνθρωποι να αντιδράσουν, η ε, οικονομική ανάπτυξη που είναι υποφελής για όλους, προσπάθειες για να προστατεύσουμε το περιβάλλον, ίσα δικαιώματα για όλους ε, και αξιοπρεπής σταθερότητα στην οικονομική ανάπτυξη για την πρώτη φορά στην ιστορία βλέπουμε ότι οι ανθρώπινες δραστηριότητες επηρεάζουν το φυσικό κύκλο του πλανήτη μας εάν συνεχίσουμε ακολουθώντας την ίδια άγουσα. Για την επόμενη γενιά θα έχουμε πάρα πολύ μεγάλες κλίμακες επιπτώσεις ε, και η μαζική φτώχεια υπονομεύει τις προσπάθειες που κάνουμε για να επιτύχουμε βιώσιμη ανάπτυξη. Αυτό είναι ένα θέμα που ενδιαφέρει τους πάντες. Θα ήθελα να τονίσω ένα πάρα πολύ σημαντικό σημείο επί του οποίου πρέπει να επιμείνουμε. Γενικώ γίνεται αποδεκτό ότι για πρώτη φορά ο κόσμος ε, έχει την τεχνολογία και τους απαιτούμενους πόρους για να εκριζώσει την ακραία φτώχεια κατά τη διάρκεια της δικής μας ζωής. Τι σημαίνει αυτό. Μέχρι το 2030 δεν θα ζήσω και πολύ με αυτά που λέω, τέλος πάντων αλλά θα πρέπει να είναι η δεδηλωμένη μας πρόθεση ότι αυτό επιδιώκουμε. Για να υλοποιηθεί το όραμα θα, ε, χρησιμοποιούμε, θα χρησιμοποιήσουμε ένα καθολικό και συνολικό πλαίσιο για την περίοδο μετά το 2015. Ένα ενιαίο σετ κανόνων που θα εφαρμόζονται σε όλες τις χώρες, λαμβάνοντας υπόψη ταυτόχρονα και τις εθνικές ιδιαιτερότητες. Γι' αυτό το φιλόδοξο θεματολόγιο χρειαζόμαστε ουσιαστικέ εταιρικέ σχέσεις που συνδυάζουν τις προσπάθειες ολονών, εθνικές κυβερνήσεις, διεθνείς οργανώσεις, διεθνή κοινότητα και τον ιδιωτικό τομέα, γιατί όχι. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη-μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο προς μεγάλη μου χαρά ε, έχουν συμφωνήσει για την πλειοψηφία των σημείων και αυτό θα αποτελέσει και τον πυρήνα αυτό του ηχηρού μηνύματος που θα περάσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην 9 Υόρκη την επόμενη εβδομάδα και έχει πραγματική υποστήριξη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο. Έχουμε την έκθεση του υψηλού πάνελ για το, την αναπτυξιακή ατζέντα μετά το 2015. Ο Γενικό Γραμματέα Σεβέν Κιμούν στην έκθεσή του ε, απηχεί αυτέ τι προτεραιότητε που υποδεικνύει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρώτη συζητήσει που έγιναν στην ομάδα εργασία για τη βιώσιμη ανάπτυξη και σχετικούς στόχους. Επίσης ε, συζήτησαν όλα αυτά τα επιμέρου σημεία, αλλά ας μην αυταπατώμεθα για να καταλήξουμε σε μια παγκόσμια συμφωνία για το πλαίσιο μετά το 2015 θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε πάρα πολύ σημαντικέ προκλήσει. και αυτό προποθέτει ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι θα ε, ε, εργαστούν με αφοσίωση γι' αυτό. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι επίσημη συμφωνία, συμφωνία συγγνώμη, μέχρι το 2015 που θα καλύπτει όλες αυτές τις και προσδιορισμό ενό οδικού χάρτη για να εξασφαλίσουμε ευημερία για όλου. Είμαι αποφασισμένος η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει ηγετικό ρόλο ε, στον παγκόσμιο διάλογο για τον προσδιορισμό τη αναπτυξιακή ατζέντα για τα επόμενα δύο χρόνια. Εμείς θα είμαστε ο συνδετικός κρίκος, θα γεφυρώσουμε το χάσμα ανάμεσα στου εταίρου, την Αφρική, του δωρητέ τον ΟΗΕ που ε, είναι ε, ένα νομιμοποιημένο βήμα προς διορισμού ε, του παγκοσμίου αναπτυξιακού θεματολογίου και επίσης για να αναπτύξουμε τις εταιρικές σχέσεις με τις αναπτυσσόμενες χώρες και την ενίσχυση τη δέσμευσή μας για την ευβιώσιμη ανάπτυξη, για την επίτευξη των στόχων του 2020 και για τη στρατηγική της πράσινης ανάπτυξης είναι μοναδική η ευκαιρία που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει το ρόλο της. Ε, στη συνέχεια ε, εννέα βουλευτέ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα ασχοληθούν επισταμένα με το ζήτημα και αυτό είναι μεγάλη προστιθέμενη αξία για να υλοποιήσουμε το πολιτικό μας όραμα. Ε, σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας. Κυρίες και κύριοι, θα είναι μεγάλη πρόκληση για να επιτευχθεί αυτό το σχέδιο για τα επόμενα χρόνια θα εργαστούμε σκληρά, αλλά όπως είπε και το πάνελ υψηλού επίπεδου, έχουμε πολύ καλή βάση. Ε, Σήμερα γίνεται και στο Παρίσι συνεδρίαση της συντακτική συνέλευση που επίση ασχολείται με αυτό το ζήτημα ε, το, της αναπτυξιακής ατζέντα και Χαρήκαμε ιδιαίτερα από την αναγνώριση που προσέφεραν οι δύο μας ε, δεν αποκλείστηκε κανείς από τη διαδικασία αυτή τη φορά. Η κοινωνία των πολιτών επίσης θεωρεί ότι μετήχε στη διαβούλευση, ακούστηκε η φωνή της. Ε, και πιστεύω ότι αυτό το άνοιγμα, η μελλοντοστραφής ε, πολιτική είναι κάτι που χρειαζόμαστε για να έχουμε ένα όχι μόνο πολιτικά ισχυρό μήνυμα αλλά να λειτουργήσει και ως όργανο για τη δράση και για την λόγοδοσία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω τώρα το λόγο στον Επίτροπο Ποτότσινικ πάλι για οκτώ λεπτά. Α, κυρίες και κύριοι αξιότιμα μέλη και των δύο επιτροπών θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την διοργάνωση αυτή της συνάντησης των, των δύο επιτροπών και θα προσπαθήσω να αναφέρω ορισμένα θέματα τα οποία νομίζω ότι θα μας απασχολήσουν όλους το μέλλον ακόμη περισσότερο. Πρώτα πρώτα να πω ότι χάρηκα που είμαι εδώ με τον συνάδελφο Πίμπελξ. Όταν έμαθα ότι θα μίλαγε πρώτα εκείνος και μετά εγώ αποφάσισα να αλλάξω τελικά την ομιλία μου για να μην επαναλάβω τα πράγματα που θα έλεγε εκείνος. Ε, Επίσης έχουμε μαζί μας και την Αμίνα... την ειδική σύμβουλο του Γενικού Γραμματέα του ΟΙΕ... η οποία θα πει παρόμοια πράγματα. Κυρίες και κύριοι, ο κόσμος τα τελευταία χρόνια έκανε αρκετή πρόοδο στον αγώνα κατά της ένδυας, αλλά δεν κατάφερε να επιλύσει το πρόβλημα. Και εκτός από την εκρίζωση της ε, ένδυας ε, άλλος μεγάλος στόχος είναι η βιώσιμη ανάπτυξη όπως έδειξαν οι συνδιασκέψεις του Γιωχάννεσμπουργκ και του Ρίο ε, υπάρχουν πολλές προκλήσεις στο μέλλον ε, για όλους μας δύο τρίτα των πόρων που χρησιμοποιούμε προέρχονται από την ίδια τη φύση, το πόσιμο νερό, το ε, φυσική πόρ, φυσικός πλούτος, πόροι κτλ. από την άλλη μεριά όμως υπάρχουν και κάποια αρνητικά από τη φύση. Οι φυσικές καταστροφές. Από το 92, οι φυσικές καταστροφές σκότωσαν πολύ κόσμο και κόστισαν πολλά χρήματα. Πολλές φορές όμως να έχουμε υπόψη μας ότι ε, υπάρχει ανθρώπινο χέρι πίσω από αυτές τις φυσικές καταστροφές και θα μπορούσαμε ίσως να αποφύγουμε κάποιες φυσικές καταστροφές αν απλώς σεβόμαστε τα όρια του πλανήτη μας. Εν πάση περιπτώσει κυρίες και κύριοι <coughs> τα προβλήματα του περιβάλλοντος, το φυσικό φαινομένων και καταστροφών και το φαινόμενο της φτώχειας ε, κάπου συνδέονται. Ε, δεν μπορούμε να... <clears throat> Δεν αρκεί μάλλον να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της μεν χώρια από τις δε. Μόνο αν δούμε τα πράγματα από κοινού μπορούμε μέχρι το 2030 να έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση που όπου μπορούμε να μιλούμε για ένα βιώσιμο μέλλον. Πρέπει να εφαρμόσουμε τις δεσμεύσεις που αναλήφθησαν πέρσι στο Ρίο τότε αποφασίστηκε ότι πρέπει να ενισχύσουμε το πλαίσιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Πρώτα-πρώτα είπαμε ότι θέλουμε να φτιάξουμε ένα ε, υψηλού επίπεδου φόρουμ για τη συζήτηση όλων αυτών των θεμάτων και εγώ είμαι πεπισμένος ότι επειδή αποφασίστηκε καταλήξαμε σε συμφωνία στο, σε οργανωτικό επίπεδο θα μπορέσουμε να ε, αντιμετωπίσουμε καλύτερα τις τρεις διαστάσεις της βιώσιμης ανάπτυξης. Περιμέν, αναμένω να μπορέσουμε να διατηρήσουμε παντού και σε όλα τα επίπεδα υψηλά στη, στην κλίμακα προτεραιότητα, στη βιώσιμη ανάπτυξη και μάλιστα σε διεθνές επίπεδο. Και επειδή είπαμε η βιώσιμη ανάπτυξη και η ακρίζωση της φτώχειας ε, συνδέονται άρρηκτα ε, οι παράγοντες ή τα μέσα που σχετίζονται ε, με τη βιώσιμη ανάπτυξη με το περιβάλλον έχουν σημαντικότερο ρόλο να παίξουν στον αγώνα κατά της φτώχειας. Η πράσινη οικονομία ε, μπορεί να βοηθήσει, είναι ένα μονοτόπιο πάτη για να καταλήξουμε στην εκρίζωση της ένδειας. Η πράσινη οικονομία είναι πολύ σημαντικό εργαλείο κατά την άποψή μου α, α, ένα απαραίτητο εργαλείο θα πρέπει να ε, προωθήσουμε την Ευρώπη 2020 ε, και να προωθήσουμε τι πολιτικές που μας οδηγούν στην πράσινη ανάπτυξη τελευταία ανάλυση. Νομίζω ότι βεβαίως αυτό το κάνουμε στο εσωτερικό της Ευρώπης είναι ευρωπαϊκά προγράμματα αυτά αλλά τα αντίστοιχα θα πρέπει να προωθούμε και σε παγκόσμιο επίπεδο όλες οι χώρες του πλανήτη θα πρέπει να προωθούν αντίστοιχες πολιτικές είναι σαφές ότι βεβαίως για τα επόμενα βήματα χρειαζόμαστε κοινή ευρωπαϊκή θέση για, τις, για να ε, συζητήσουμε σε διεθνές επίπεδο. Και εδώ πραγματικά νομίζω ότι είναι τρία τα σημαντικά θέματα. Πρώτο, στόχοι για την βιώσιμη ανάπτυξη θα πρέπει να εφαρμόζονται καθολικά. Είναι ένα όραμα για το μέλλον όπου πρέπει να εμπλακούν όλοι οι φορείς, όλες οι χώρες. Δεν πρόκειται για μία ατζέντα μόνο για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Για όλες τις χώρες, τις αναπτυγμένες, τις αναπτυσσόμενες, τις νέες οικονομίες, για όλους. Θέλουμε όλοι να αναλάμβουν ε, δεσμεύσεις σχετικά με βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση. Δεύτερο θέμα, όταν αναπτύσσουμε τους καινούριου στόχους θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η, οικονομ... η... η... ότι η βιώσιμη ανάπτυξη δεν ξεχωρίζει ανάμεσα στην στον οικονομικό τομέα, στον κοινωνικό τομέα κτλ. Πρέπει να δημιουργήσουμε διασυνδέσεις, παραδείγματος χάρη, ε, μεταξύ ε, ποιότητας του αέρα και υγείας, μεταξύ νερού και γης, μεταξύ νερού, γης και ενέργειας. Αυτά όλα συνδέονται και πιστεύουμε ότι αν βρούμε λύσεις για όλα αυτά που μας απασχολούν σχετικά ε, μοιραία βοηθούμε και στην εκρίζωση της φτώχειας. Επίσης τέλος θα πρέπει οι στόχοι μας ε, θα πρέπει οι στόχοι να βασίζονται και σε δείκτες επιστημονικούς, ε, ερευνητικούς και η σχέση μας με το, όλους τους ενδιαφερόμενους να είναι φύση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συνεργαστεί με όλους εκείνους που ενδιαφέρονται, με όλους αυτούς που α, πονάνε τον πλανήτη. Όπως είπε και ο πρόεδρος Μπαρόζο, μέχρι το τέλος της θητείας μας θα συνεχίσουμε να επιμένουμε στους στόχους της χιλιετίας για να μπορέ... και στους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης και αν θέλουμε πραγματικά να επηρεάσουμε σημαντικά τον διεθνή διάλογο θα πρέπει ήδη από τις αρχές της επόμενης χρονιάς να έχουμε ε, οριοθετήσει το τι θα κάνουμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να μπορέσει να δράσει σαν ανοιχτός και αποτελεσματικός διαπραγματευτικός εταίρος μέχρι την Σύνοδο Κορυφής του 2015. για τις πρωτοβουλίες που πήραν και οι δυο επιτροπές για τα θέματα μετά το 2015 και ευχαριστούμε εκ των προτέρων όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πιστεύουμε ότι θα μας βοηθήσουν να ε, διατηρήσουμε την ορμή και να επιτύχουμε τους στόχους μας. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα ακούσουμε την ειδική σύμβουλο Αμίνα Μοχάμετ για 8 λεπτά. Ευχαριστώ, αξιότιμοι πρόεδροι, αξιότιμοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι. Με τιμά η παρουσία μου εδώ σήμερα. Μου δώσατε την ευκαιρία να μιλήσω ενώπιον σε αυτή τη μεικτή συνεδρίαση των Επιτροπών ΔΕΒΕ και ΕΜΒΗ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους ιδιαίτερους πρόεδρους των δύο Επιτροπών για αυτή την πρόσκληση. Η στόχη της χιλιετίας είναι βασική καμπή ε, στο να ε, ενισχύσουμε την πολιτική βούληση για ανάληψη αυτής δράσης και έχει σημειωθεί συγκεκριμένη πρόοδος, όμως ε, ε, ε, υπάρχουν μεγάλες διαφορές ανάμεσα στα κράτη και τις περιοχές. Επάνω από ένα δις άνθρωποι ζουν σε ακραία φτώχεια και υπερβολικά μεγάλο ποσοστό έχουν σοβαρές ελλείψεις ως προς την παιδεία και τις υπηρεσίες υγείας και διευρύνεται το χάσμα ανάμεσα στα φύλλα, το εισόδημα, την εθνότητα, την ηλικία, τον τόπο διαμονής. Όσο προσεγγίζουμε το 2015 η διεθνής κοινότητα επιταχύνει τις προσπάθειές της για την υλοποίηση των των στόχων. Η επίτευξη αυτών των στόχων θα πρέπει να παραμείνει ύψιστη προτεραιότητα για μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο και να ζητήσω ε, και από το Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη αρρωγή για την επίτευξη των στόχων της χιλιετίας, διότι η αξιοπιστία του επόμενου θεματολογίου θα είναι συνάρτηση της επιτυχίας του προηγουμένου. Ε, και ακόμη και αν ε, επιτευχθούν οι στόχοι της χιλιετίας ε, υπολείπεται μεγάλο έργο και εξάλλου έχουν προκύψει και νέες σημαντικές προκλήσεις. Έχει διωγγωθεί η ανισότητα, η έλλειψη πόρων υπονομεύοντας το μέλλον μας. Πλέον κανείς δεν αμφισβητεί τις επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών και όλοι ζητούν ανά τον κόσμο πιο υπεύθυνη διακυβέρνηση και αυτό σε όλα τα επίπεδα. Η μετανάστευση και το θέμα της υπερβολικής αστυνομίας ε, δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα. Ε, ε, κάποιες χώρες έχουν πλέον, ακολουθούν μια αντίστροφη πορεία λόγω ενόπλων σειράξεων και πλήττονται περισσότερο οι γυναίκες και τα παιδιά. Ως προς το λαθρεμπόριο των ναρκωτικών βλέπουμε σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τώρα χρειαζόμαστε μια παγκόσμια ατζέντα για να καλύψουμε όλες αυτές τις ανησυχίες, αλλά ξαναλέω ύψιστη προτεραιότητα πρέπει να είναι η εκρίζωση της φτώχειας ταυτόχρονα να πρέπει να κλιμακώσουμε τις προσπάθειε μας για να επιτύχουμε μια νέα δυναμική για την βιώσιμη ανάπτυξη και μια ανάπτυξη με χαμηλή, ε, χαμηλές εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Ε, γίνονται όλο ένα και πιο διατομιακές, ε, διαγενειακές ε, οι προκλήσεις. Ε, ο ΙΕ τον περασμένο χρόνο έχει κάνει μία σειρά διαβουλεύσεις σε πάρα πολλά επίπεδα. Είναι ευρύτατο φάσμα που ε, καλύπτει ε, πάρα πολύ μεγάλο αριθμό περιοχών ανά τον κόσμο. Μπορέσαμε να ακούσουμε τη φωνή εκατομμυρίων ανθρώπων για το θεματολόγιο μετά το 2015 για να προσδιορίσουμε τον κόσμο που θα ήθελαν να δημιουργηθεί. Γιατί το επόμενο θεματολόγιο πρέπει να έχουμε υπόψη υπόψη ότι και οι προηγούμενε και οι τωρινέ προκλήσει ε, ε, συνεπάγονται βασικέ αλλαγέ, ε, όχι μόνο ω προ τι αρχέ, αλλά και τον τρόπο λειτουργία που ακολουθεί η διεθνή κοινότητα. Είναι ακόμη πρόωρο για να προδικάσουμε την έκβαση των διαβουλεύσεων ε, που θα γίνουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας για τον προσδιορισμό της Ατζέντα 2015. Παρ' όλα αυτά ξέρουμε ότι η οικονομική ανάπτυξη, η κοινωνική ένταξη και η περιβαλλοντική βιωσιμότητα είναι τρεις βασικές αρχές που θα στηρίξουν αυτή την αλλαγή των αρχών ε, και του τρόπου ε, δράσης που αναλαμβάνουν τα κράτη-μέλη. Είναι μοναδική ευκαιρία που έχουμε για να ενσωματώσουμε αυτές τις τρεις συνιστώσεις σε μια σφαιρική προσέγγιση έχοντας την ανάπτυξη στον πυρήνα του επόμενου θεματολογίου τόσο ώστε να καλύψουμε τις πραγματικές ανάγκες και επιθυμίες των ανθρώπων. Χρειαζόμαστε λοιπόν κοινή προσέγγιση για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις και η βιώσιμη ανάπτυξη είναι το μοναδικό μονοπάτι, ο μονόδρομος του μέλλοντος. Ε, επιταχύνεται η πρόοδος για την επίτευξη των στόχων της χιλίτιας και ο σχεδιασμός ε, έχει ε, σημασία που δεν μπορεί να υποτιμηθεί. Είναι τεράστια μεγάλης κλίμακας και χρειαζόμαστε σχεδιασμό και επίσης αυτό που χρειάζεται να κάνουμε είναι να ακούσουμε τη φωνή των ανθρώπων και γι' αυτό το Κοινοβούλιο έχει κέριο ρόλο να διαδραματίσει σε αυτή τη διαδικασία. Κυρίε και κύριοι, πριν από ένα χρόνο δεν θα ήμουν ε, τόσο αισιόδοξη όμω. Τώρα ε, είμαι πεπισμένη ότι ακολουθεί τη σωστή κατεύθυνση η διεθνή ε, κοινότητα για το σχεδιασμό για την περίοδο μετά το 2015 και μπορώ να ευχαριστήσω και τον Αντρέ και τον Γιάννη. Γι' αυτό εργαστήκαμε πάρα πολύ σκληρά, ούτω ώστε να ενώσουμε τα δύο θεματολόγια και να καταλήξουμε σε μια κοινή προσπάθεια. Ε, τώρα είναι πλέον πλήρως λειτουργικά ε, τα αποτελέσματα, τα συμπεράσματα της ομάδας εργασίας. Έχουμε τη Διακυβερνητική Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων για τη Βιώσιμη Χρηματοδότηση, η οποία θα ολοκληρώσει μέχρι το Σεπτέμβριο του 2014 τις εργασίες της. Επίσης, το Πολιτικό Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου, που θα δρομολογηθεί στις 24 Σεπτεμβρίου, αναμένεται να εργαστεί με πολύ αποτελεσματικό τρόπο. Εκατομμύρια ανθρώπων ακούστηκαν σε αυτές τις άνευ προηγουμένου παγκοσμίου κλίμακας διαβουλεύσεις. Ένα εκατομμύριο φωνές, λοιπόν, λοιπόν. Τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων δημοσιεύθηκαν την περασμένη εβδομάδα. Ε, για το, την ατζέντα του 2015 βλέπουμε ότι οι κλιματικές αλλαγές είναι βασική απειλή για την αξιοπρεπή διαβίωση, για την ειρήνη, την ασφάλεια και επηρεάζει τη ζωή μας με πολλούς τρόπους. Για να αντιμετωπίσουμε τις κλιματικές αλλαγές ε, χρειάζονται δράσεις που ταυτίζονται με τις δράσεις που χρειαζόμαστε για την εκρίζωση της στόχης και εντόνωση της ανάπτυξης. Έχουμε βεβαίως διαφορετικές ε, ε, κυβερνήσεις κυβερνητικές ε, μεθόδους, ε, όμως ε, θα πρέπει να αντιληφθούμε πώς διασυνδέονται, ούτω ώστε να εξασφαλίσουμε ότι θα καταλήξουμε σε μέτρα που αλληλοσυμπληρώνονται και όχι επικαλύπτονται. Η έκθεση του Γενικού Γραμματέα, μια αξιοπρεπή διαβίωση για όλους, περιγράφει το όραμα του Γενικού Γραμματέα για την περίοδο μετά το 2015 και συμπεριλαμβάνει βασικές συστάσεις προς τα κράτη-μέλη που θα πρέπει να συνεκτιμηθούν κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Βλέπουμε συνένεση για ένα παγκόσμιο θεματολόγιο, ένα θεματολόγιο που θα εφαρμόζεται σε όλες τις χώρε, και κανείς δεν θα αποκλείεται από αυτή τη διαδικασία. Η βιώσιμη ανάπτυξη είναι στον πυρήνα και η βασική αρχή, ξαναλέω, είναι η εκρίζωση της στόχιας, είναι στην προτεραιότητα ε, και η ε, ε, οι περιβαλλοντικές ανησυχίες και οι οικονομικές ανησυχίες είναι αυτές που θα διέπουν την διαδικασία. Εξάλλου που συμφωνήθηκε στην διάσκεψη Ρίο Συνήκωση. Επίσης το κράτος δικαίου, οι θεσμοί, η σχέση ανάμεσα στην ανάπτυξη και η ειρήνη νομίζω είναι αυτονόητη για όλους και αυτό δεν εφαρμόζεται μόνο σε μια παγκόσμια εταιρική σχέση αλλά και σε επίπεδο κρατών μελών ε, για να ληφθούν υπόψη οι τοπικέ ε, ε, προτεραιότητε, Χρειαζόμαστε ένα διεθνέ σύστημα όπου θα μετάσχει ο ΙΕ για να έχουμε μια συντονισμένη απόκριση και να επιτύχουμε του στόχου μα. Επίση, ισχυρό σύστημα εποπτείας και παρακολούθηση. Αυτό έχει κέρια σημασία για την παρακολούθηση τη εφαρμογή του δηματολογίου μετά το 2015 και εκεί είναι κεντρικό ο των κυβερνήσεων των κρατών μελών. Μπορούμε να ενισχύσουμε την εποπτεία αν εμπλάκουν άμεσα και οι πολίτε καθώ και οι μικρέ επιχειρήσει, ε, ούτω ώστε να χρησιμοποιηθούν και οι νέε τεχνολογίε ε, για να αποομαδοποιήσουμε δεδομένα και να μειώσουμε το κόστο συλλογή ε, των δεδομένων. Νομίζω ότι έχουμε βρει τα πιο, το πιο πρόσφορο τρόπο δράση και η διεθνή κοινότητα έχει τι απαιτούμενε οργανώσει και του μηχανισμού για να μπορέσει να καλύψει καταλήξει σε ένα παγκόσμιο θεματολόγιο που θα μπορέσει να εφαρμοστεί και στο τοπικό επίπεδο. Υπάρχουν αλληλοσυνδεόμενε προκλήσει. χρειαζόμαστε πραγματική οικονομική μεταμόρφωση του κόσμου και μια νέα ε, παγκόσμια εταιρική σχέση ε, χρειαζόμαστε όμως ταυτόχρονα και συνοχή και αποτελεσματικότητα για τον οδικό χάρτη μετά το 2015. Είναι ιδιαίτερα περίπλοκες διακυβερνητικές διαδικασίες. Ε, τώρα, οι ειδικέ εκδηλώσεις ε, που θα γίνουν στις 25 ε, υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα θα ανοίξουν το δρόμο για να αρχίσουν οι διαβουλεύσεις για το θεματολόγιο μετά το 2015 ε, για την επίτευξη των στόχων ε, της χιλιετίας αλλά και για να υπάρξει πολιτική συσπήρωση για την επιτάχυνση της δράσης μας. Ε, Αντιλαμβανόμαστε ότι η Ιρλανδία λαμβάνει ηγετικό ρόλο διότι συμπροεδρεύει στο δεύτερο ήμιση του 2013 και το σύστημα του ΕΕ από, ε, ε, από μια διαβουλευτική φάση περνάει σε μια φάση όπου επιδιώκει την εξέβρεση συνένεσης. Ε, Στου επόμενους 12 μήνες ε, η ομάδα εργασίας για τους στόχους χιλιοετίας, το πολιτικό φόρουμ υψηλού επίπεδου, η Επιτροπή Έμπειρο Γνωμόνων για τα χρηματοπιστωτικά το Σεπτέμβρη θα καταθέσουν τα συμπεράσματά του για να ξεκινήσει και τελική φάση των διακυβερνητικών διαβουλεύσεων στα πλαίσια τη γενική συνέλευση. Ε, είναι πραγματικά μεγάλη πρόκληση και ε, ιστορικού χαρακτήρα για τα κράτη-μέλη ε, του ΟΗΕ. Ξέρετε ότι δεν θέλουμε να αποκλειστεί κανεί από αυτή τη διαδικασία που θα καθορίσει τον μέλλον μα Είναι καταπήγον το ζήτημα και γι' αυτό η Διεθνή κοινότητα πρέπει να υπερβεί τα γεωπολιτικέ και ιδεολογικέ διαιρέσει, ούτω ώστε να είναι φιλόδοξη φιλόδοξη, φιλόδοξο το νέο θεματολόγιο που θα οικοδομεί. Σα ευχαριστούμε για την οικοδομητική σα συμμετοχή σε αυτή τη διακυβερνητική ε, διαδικασία διαβουλεύσεων στη Νέα Υόρκη. Ευχαριστούμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση για την υποστήριξή του σε όλη αυτή τη διάρκεια διαβουλεύσεων πολλαπλών επιπέδων. Ξαναείπαμε ε, στο πολιτικό πάνελ υψηλού επίπεδου, ε, η Task Team του ΟΗΕ, το δίκτυο των βιώσιμων λύσεων και το Παγκόσμιο Σύμφωνο για τις επιχειρήσεις. Επίσης, ευχαριστούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, για την ε, προσπαθεί και επιδιώκει ένα σφαιρικό θεματολόγιο και όχι μια τμηματική προσέγγιση. Ε, αυτό ε, επαναλήφθηκε στις περάσματα του τελευταίου Συμβουλίου στο Λουξεμβούργο και θα θέλουμε να συγχαρούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτή την εξέλιξη. Ελπίζουμε ότι αυτό, αυτή η νέα προσπάθεια θα τροφοδοτηθεί και θα μας βοηθήσει να υπερβούμε αυτόν τον εθνικό καταγερματισμό ή τον τομεακό, τον υπηρεσιακό και καταγερματισμό για να εργαστούν όλοι για την επίτευξη κοινών στόχων. Ο ρόλο σας είναι κύρια σημασία γιατί πρέπει να καθοδηγήσετε το διεθνή κοινότητα ώστε να καταλήξει σε μία ενιαία συνεκτική ατζέντα μετά το 2015. Εν κατακλείδη εξοχότες κυρίες και κύριοι θα ήθελα να πω ότι είμαστε η πρώτη γενιά που έχει τους πόρους και την πραγματογνωμοσύνη για να θέσουμε ένα, ε, θέσουμε ένα τέρμα στην ακραία φτώχεια και να τονώσουμε, να επιτύχουμε την βιώσιμη ανάπτυξη. Προτού είναι αργά. Ε, συνεχίζονται οι όχι μόνο στην Νέα Υόρκη αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο για τα ε, βασικά ζητήματα, ε, τη χρηματοδότηση, την καθολικότητα του ε, προγράμματο διαφοροποίηση ω προ το σχεδιασμό και τις ευθύνε, και επίση ο τρόπος παραγωγής, επιταγή δηλαδή της ατζέντα για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Νομίζω ότι έχουμε μια καταπληκτική ευκαιρία για να επιδιώξουμε την επίτευξη αυτών των στόχων. Ελπίζω όλοι να συσπηρωθούμε για να καταλήξουμε καταλήξουμε σε ένα συνολικό πλαίσιο για μετά το 2015, έχοντα ξαναλέω βασική προτεραιότητα την εκρίζωση τη φτώχεια και τι οικονομικέ ευκαιρίε για όλου. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αξιοποιήσουν αυτή τη μοναδική ευκαιρία και πρέπει να συνεργαστούμε όλοι για να οικοδομήσουμε ένα καλύτερο κόσμο που όλοι θα ζουν αξιοπρεπώ και θα έχουν καλύτερο δυναμικό. Η μεγαλύτερη πρόκληση να μην αποκλειστεί κανεί. Πρέπει να του πρόξουμε όλου προ τα μπροστά. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σα. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στους συναδέλφους μου. Θα ξεκινήσω με τον κύριο Κάτσμαρεκ. Όχι, για μια στιγμή. Για δυόμιση λεπτά κύριε Κάτσμαρεκ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε μάλλον, κυρίες και κύριοι. Συμφωνώ απολύτως με αυτά τα οποία μας είπε και ο Επίτροπος Πίμπαλξ. Πράγματι σήμερα μπορεί κανείς να είναι σχετικά πιο αισιόδοξο για την επίτευξη των στόχων της χιλιετίας. Το 2004 όταν πήρα για πρώτη φορά μέρος της εργασίας μας ήμουνα πολύ πιο διστακτικός. Και παρά το ότι ζούμε μια περίοδο κρίσης οικονομική μπορούμε να είμαστε πιο αισιόδοξοι. Γιατί αυτό. Ίσως γιατί υπάρχει καλύτερης καλύτερος συντονισμός, ίσως γιατί με το χρόνο έχουμε αποκτήσει εμπειρία, πάντως είμαστε πολύ πιο κοντά στην ουσιαστική επίτευξη των στόχων της χιλιετίας από ό,τι πριν λίγο καιρό. Δεύτερον, θα ήθελα να πω, υπάρχει μια μεγάλη συνένεση ανάμεσα στην Επιτροπή και το Κοινοβούλιο και σε επίπεδο συμβατότητας των εγγράφων μας της ανακοίνωσης δηλαδή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της εκθέσεως που οποία, την οποία υιοθετήσαμε αλλά και ε, στρατηγική συμφωνία για τους στόχους τους οποίους επιδιώκουμε. Οι στρατηγικοί αυτοί στόχοι θα πρέπει να υιοθετηθούν θα έλεγα από κοινού. Απαιτείται να είμαστε ε, μαζί, φιλόδοξοι και να προσπαθήσουμε να μετρήσουμε σωστά τους στόχους αυτούς κατά προτεραιότητα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το έχει ήδη πει και το, και το Κοινοβούλιο το έχει ήδη πει. Υπάρχει σύμπτωση απόψεων ανάμεσα στα δύο όργανα. Η πρόεδρος μας το υπογράμμισε. Θα πρέπει να εντάξουμε και την αηφόρο ανάπτυξη και την προστασία του ε, περιβάλλοντος. Εάν πράγματι ολοκληρώσουμε σε μία προσπάθεια τα δύο αυτά στοιχεία, τότε θα υπάρχει η πιθανότητα να μην κάνουμε τα ίδια λάθη τα οποία έχουν γίνει σε χώρες οι οποίες σήμερα είναι αναπτυγμένες, αλλά των οποίων οι μορφές ανάπτυξης δεν ήταν αηφόρες και το τίμημα το πληρώνουν σήμερα όλοι και οι αναπτυγμένες και οι σε ανάπτυξη χώρες. Αν καταφέρουμε να συνδυάσουμε λοιπόν το στοιχείο της αηφορίας και το στοιχείο του σεβασμού του περιβάλλοντος, τότε θα μπορέσουμε ίσως να μην ξανακάνουμε το ίδιο λάθος για δεύτερη φορά. Ακολουθούμε λοιπόν διαφορετικές πορείες και έχουμε διαφορετικούς στόχους, αλλά παρόλα αυτά είναι φυσιολογικό να υπάρχει θα έλεγα μία σύγκρουση ανάμεσα σε αυτά τα μέσα τα οποία λειτουργούν ανταγωνιστικά το ένα με το άλλο και αντί να πετύχουμε τους στόχους ξεκινάμε συζητήσεις, στήρες για το ποιες είναι οι πιο σημαντικές από τις προσπάθειες που πρέπει να γίνουν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Κάσμαρεκ. Ο κύριος Κάσμαν έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε να ευχαριστήσω τους εκλεκτούς προσκεκλημένους. Δεν, συμφωνώ, ε, δεν διαφωνώ καθόλου με αυτά τα οποία είπατε, αλλά έχοντας διαβάσει προσεκτικά τα διάφορα εγγραφά και την έκθεση του πάνελ επίπεδου, δεν υπάρχει καμία αναφορά στις λεσβίες, στους ομοφιλόφιλους άνδρες, γυναίκες κτλ. Εκτός από μία αναφορά στις, ε, στις στο τέλος. Χαίρομαι που υπάρχει αναφορά στις γυναίκες, αλλά πώς μπορεί κανείς να πετύχει τους στόχους του ε, εμείς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, δίνουμε μάχες με τους συναδέλφους ε, των ΑΚΕ για τα βασικά δικαιώματα των ομοφιλόφιλων ανδρών και γυναικών. Πώς μπορούμε εμείς να πετύχουμε την ισοτιμία μπροστά στον νόμο και την δίκαιη προστασία. Νομίζω ότι οι προσπάθειες που έχουν γίνει τώρα για την προώθηση των δικαιωμάτων όλων είναι κάτι που δεν πρέπει να το αγνοούμε. Υπάρχει μία λέξη λοιπόν που συμπεριλαμβάνει όλους τους ανθρώπους σε αυτό τον πλανήτη. Όλοι. Αν δεν βάλουμε την ε, λέξη όλοι, αυτό σημαίνει ότι και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε επίπεδο ε, Ηνωμένων Εθνών μια ιεραρχία των δικαιούχων προστασίας και αυτό είναι απαράδεκτο. Η κυρία Γκρέζ, ευχαριστώ πρόεδρε. Είναι αλήθεια ότι η πιο σημαντική συνάντηση οδήγησε στη δήλωση της χιλιετίας. Πού βρισκόμαστε τώρα. Ε, βλέπουμε ότι δεν έχουμε πετύχει πολλούς στόχους, βλέπουμε ότι υπάρχει μια χειροτέρευση των δικαιωμάτων. Ο κύριος Κάσμαν είπε ότι δεν έχουμε ρυθμίσει το θέμα των δικαιωμάτων αυτών που έχουν, ε, θα έλεγα, σεξουαλικούς ε, προσδιορισμούς και προσανατολισμούς διαφορετικούς. 1,3 δις ανθρώπων στον πλανήτη ζούνε με κάτω από ένα ευρώ την ημέρα. Η διαφθορά κυριαρχεί, τα προβλήματα ε, τα σχολικής εκπαίδευσης παραμένουν. Γενικά και οι συγκρούσεις συνεχώς χαίνουν. Συνεπώς λοιπόν ναι μεν έχουμε ψηφίσει κάποιους στόχους ε, της χιλιετίας για την ανάπτυξη και επί τη βάση του κυρίου, της προτάσεως του κυρίου Κάτσμαρεκ που είχε προτείνει να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια, περισσότερα ανθρώπινα δικαιώματα και σωστή χρηστή διακυβέρνηση. Άλλωστε και μια ομάδα υψηλού επίπεδου ε, λειτουργήσε ε, σωστά. Πάντως θα ήθελα να πω ότι αν δεν καταπολεμήσουμε αποτελεσματικά την φοροδιαφυγή, την νομιμοποίηση παράνομου χρήματος. Αν δεν προχωρήσουμε στην αποκατάσταση των εμπορικών σχέσεων με ισόρροπο τρόπο, τότε δεν θα πετύχουμε τους στόχους μας. Θα πρέπει λοιπόν να θέσουμε ένα τέλος στις ανισότητες, στις κρίσεις στην αντιμετώπιση των προβλημάτων ε, στη συνέχεια των κλιματολογικών αλλαγών, στην απώλεια της βιοπικιλότητας, απαιτείται μια ουσιαστική ριζοσπαστική αλλαγή στον τρόπο παραγωγής και κατανάλωσης. Δεν μπορούμε να τα αυτό. Δεν μπορούμε να κάνουμε μόνο επιμέρους ε, προσπάθειες. Χρειάζεται μια ολοκληρωμένη προσπάθεια που να λαμβάνει υπόψη και τη διάσταση την οικονομική και την κοινωνική για το σύνολο των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια, θα συμφωνήσουμε όλοι λέγοντας ότι η καταπολέμηση της φτώχειας και η αηφορία δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με διαφορετικό τρόπο. Αλλά εγώ δεν συμμερίζομαι την ισιοδοξία του Φίλιπ Κάτσμαρεκ. Νομίζω ότι έχουμε να κάνουμε με μια ουσιαστική πρόκληση. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε ένα νέο τρόπο ανάπτυξης συμβατό με τα όρια, τα περιορισμένα πλέον όρια των πόρων, των φυσικών που έχει ο πλανήτης. Εφαρμόζοντας τα πρότυπα του Βορρά στον Νότο δεν θα το πετύχουμε αυτό. Έχω και αρκετές ερωτήσεις για τους επιτρόπους. Πώς μπορούμε εμείς να βοηθήσουμε, να βοηθήσουμε την, την ενεργειακή μετάβαση ε, στο Νότο και τι συγκεκριμένες ενέργειες έχουν γίνει από την Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι ώστε η φορεία στην ανάπτυξη να είναι καθοριστική για την πολιτική αυτή. Ευχαριστώ κύριε Γκρέζ. <clears throat> Κλάις. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και ευχαριστώ για την κοινή αυτή συνεδρίαση ε, των δυο επιτροπών. Από τις ομιλίες που έγιναν έγινε σαφές και είναι πραγματικότητα ότι αγωνιζόμαστε κι εσείς και εμείς ε, όλοι μας εδώ να συγκεράσουμε τις προσπάθειές μας ε, από τους δύο τομείς τους οποίους δραστηριοποιούμε. Αναρωτιέμαι όμως αν έχουμε στη διάθεσή μας τα σωστά, τα κατάλληλα εργαλεία και θα ήθελα να δω τώρα, να θυμίσω α, αυτά που έγιναν την περασμένη εβδομάδα τη συζήτηση για τα βιοκαύσιμα. Ε, όλοι έχουμε στη διάθεσή μας τα τα κατάλληλα εργαλεία θέλουμε όλοι να διατηρήσουμε τα τροπικά δάση με τι μέσα, με τι εργαλεία πρέπει να κάνουμε ε, προσπάθειες για μια ε, κατανάλωση πιο συνειδητή ε, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να απαγορεύσουμε κάποιες τεχνικές που οδηγούν σε υπερβολική διάβρωση ε, ορισμένων περιοχών του πλανήτη που πρέπει να προστατευθούν ιδιαίτερα στα τροπικά λάθη ε, δάση και όταν λέμε τροπικά δάση δεν μπορούμε βέβαια να ξεχνάμε και το κλίμα ξέρουμε πολύ καλά ότι ε, είμαστε ότι ξέρουμε ότι μας χρειάζονται ορισμένοι πόροι γιατί πραγματικά για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε τα, τα δάση μας θα πρέπει να πληρώσουμε και το αντίτιμο. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά να τα έχουμε κατά νου. Και σας λέω όλοι πρέπει να αγωνιστούμε από κοινού. Ευχαριστώ πολύ λέει ο πρόεδρο, η πρόεδρος, ο κύριος Τουριολιά έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε, κύριε Επιτροπή. Ε, χαίρομαι που συναντιόμαστε εδώ που συναντιόμαστε λίγε, λίγο καιρό πριν από τις πολύ αποφασιστικές συζητήσεις που θα γίνουν για το μέλλον του πλανήτη. Από τη μια έχουμε τον πλανήτη και το περιβάλλον, και από την άλλη έχουμε που πρέπει να διατηρήσουμε, από την άλλη έχουμε την καταπολέμηση της ένδυας. Είναι διπλή πρόκληση και πραγματικά θέλουμε αν είναι δυνατόν να προχωρήσουμε τον ίδιο ενθουσιασμό και στα δυο. Ε, θα πρέπει να βρούμε κανονιστικές ρυθμίσεις για μετά το 2015 που να εφαρμοστούν με το σωστό τρόπο. Όταν λέει ο Επίτροπος ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλα τα, χρημα, οικονομικά μέσα που έχουμε για την περίοδο μετά το 2015 όταν ξέρουμε ότι χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί και ο δημόσιος και ο ιδιωτικό τομέας αυτό σημαίνει ότι όλοι θα πρέπει να αγωνιστούμε διότι πραγματικά ε, είναι αλήθεια ότι η βιώσιμη ανάπτυξη και η καταπολέμηση της φτώχειας συνδέονται και αν δεν τα καταφέρουμε είναι να, σαν να ανοίγουμε το κουτί της Πανδώρας και δεν ξέρουμε τι μας περιμένει. Πραγματικά πιστεύουμε και είναι πρέπει λοιπόν να ε, προσπαθήσουμε και αν η πολιτική ανάπτυξη δούμε ότι δεν αρκεί θα πρέπει να επιμείνουμε για να χρησιμοποιήσουμε ορίσουμε ε, στάνταρτ πρότυπα τα οποία να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ενδεχομένω να χρησιμοποιήσουμε και κονδύλια για την καταπολέμηση της φτώχειας για να διατηρήσουμε την ανάπτυξη. Στη Γαλλία παραδείγματος χάριν ε, γίνεται προσπάθεια τα η βιώσιμη ανάπτυξη να μπει σε όλα τα ε, έργα τα οποία οποία ε, εφαρμόζονται και υλοποιούνται. Ε, αυτό θα πρέπει να το κάνουν και οι άλλες χώρες. Ξεκινάει λοιπόν σήμερα μια ε, μεγάλη συζήτηση που ελπίζουμε να οδηγήσει σε αυτά αποτελέσματα γι' αυτό χαιρόμαστε που είμαστε μέλη αυτής της συζήτησης και τώρα ο κύριος Μίτσελ έχει το λόγο ευχαριστώ πρόεδρε Ξέρω ότι η οι στόχοι της χιλιετίας που συγκλίνουν και είναι αποτελεσματικοί είναι ίσως ευσεβείς πόθη για ορισμένους όμως όπως ε, ίσως έχω πει και στο παρελθόν ε, θα πρέπει να καθίσουμε να σκεφτούμε τη χρήση των πόρων που έχουμε στη διάθεσή μας ε. Στα, αυτή τη στιγμή ζούμε μια κρίση ε, και τα κράτη-μέλη όλα εφαρμόζουν προγράμματα λιτότητας. Οπότε θα πρέπει και εμείς να δράσουμε στο ίδιο πλαίσιο. Είναι πολύ σημαντικό να το έχουμε αυτό υπόψη μας. Και γι' αυτό θα ήθελα να ρωτήσω, να ζητήσω ε, και, και από τους δυο επιτρόπους να... Ε, να προσπαθήσουν να βάλουν στην ημερήσια διάταξη α ε, τα ποσά αυτά τα οποία εξοικονομούμε από τη μείωση των ε, κινδύνων των φυσικών καταστροφών, των, από τις καταστροφές είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι αν ότι όλοι μαζί μπορούμε. Ε, έχουμε μία έκθεση η οποία μας δείχνει ότι το κόστος της μη Ευρώπης είναι 800 εκατομμύρια το χρόνο. Θέλουμε λοιπόν και αποτελεσματικοί να είμαστε και να εξοικονομούμε. Σε τελευταία ανάλυση όμως δεν εξοικονομούμε μόνο πόρους, εξοικονομούμε ζωές. Θα πρέπει λοιπόν να ξανακαθίσουμε, να προσέξουμε τη χρήση των πόρων που έχουμε στη διάθεσή μας, των μέσων που έχουμε στα διάθεσή μας, να, να συζητούμε τα θέματα αυτά λοιπόν σε όλα τα επίπεδα και σε εθνικό και στα εθνικά κοινοβούλια και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και άλλα παρακαλώ να βάλετε και το Disaster Risk Reduction στην ημερήσια διάταξη. Ο κύριος λέει. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε αυτή τη συζήτηση σήμερα, μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Και εγώ εδώ και κάποια χρόνια, αντιμετωπίζοντας μάλιστα ορισμένα προβλήματα υγείας, αναγκάστηκα να σκεφτώ το θέμα της υγείας και πράγματι νομίζω ότι έχουμε να κάνουμε με μία έννοια η οποία συγκεντρώνει το σύνολο των λαθών τα οποία κάνουμε. Γνωρίζουμε σαν παράδειγμα εν πολύ σήμερα ότι ο καρκίνος εξακολουθεί να επηρεάζει και να αυξάνεται αρνητικά φυσικά και υπάρχουν και πάρα πολλές άλλες ασθένειες οι οποίες επίρχουν και οι οποίες ε, επιμένουν και τα συστήματα υγείας ε, δεν φαίνεται να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά. Χτες μάλιστα είχα προτείνει μια τροπολογία γύρω από το θέμα αυτό και θα ήθελα το θέμα της υγείας να είναι ένα τμήμα ε, το οποίο να αναφέρεται συγκεκριμένα σαν βασικός στόχος της ασφάλειας και της πολιτικής μας. Είναι ένα κεφάλαιο όδες θα έλεγα σημείο της προσπάθειά μας για ένα καλύτερο μέλλον. Η πολιτική για την υγεία δεν αφορά μόνο τα εισοδήματα αναπολίτη, αλλά είναι κάτι το οποίο ε, έχει σχέση και με τον τρόπο με τον οποίο ζει ο άνθρωπος και από μια σειρά ε, γενικά ε, παραγόντων που επηρεάζουν αρνητικά την υγεία και στις φτωχές κυρίως αλλά και στις πλούσιες χώρες. Πρόκειται, θα έλεγα, τα προβλήματα της υγείας στην ουσία αποτελούν ένα υπόδειγμα ε, αρνητικής επίπτωσης της φτώχειας. Πρέπει λοιπόν να δώσουμε ένα άλλο παράδειγμα, ένα παράδειγμα το οποίο να είναι συμβατό και με, τις, με τους κανόνες της ίδιας της φύσης, να προσπαθήσουμε να δώσουμε εγγυήσει για μια καλύτερη ανθρώπινη υγεία, κάτι το οποίο θα επιτρέψει ε, στους πολίτες αυτών των χωρών μας να ζήσουν καλύτερα. Την προηγούμενη εβδομάδα είχα σαν παράδειγμα την δυνατότητα να δω από κοντά το τι συμβαίνει στην Ινδία ε, έχουν κάποιες μορφές ε, ε, οικονομικής καλλιέργειας όπως λέγεται στην Ινδία είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει. Είναι ένα πάρα πολύ καλό θέμα το οποίο πρέπει να απασχολήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και η Επιτροπή και οι εκπρόσωποι των Ηνωμένων Εθνών ε, μου δημιουργούν ένα αίσθημα ε, ε, λύπης γιατί όλοι αυτοί οι στόχοι εδώ μαζεύονται ε, σε ένα και τον ίδιο κορβανά και γίνεται προσπάθεια να υλοποιηθούν όλοι μαζί. Αυτό είναι τεράστιο έργο του στο οποίο φοβάμαι ότι θα αποτύχουμε. Μέχρι τη είναι πολύ δύσκολο ε, μέχρι την επόμενη άνοιξη που θα γίνουν οι ε, ευρωεκλογές να μπορέσουμε να κάνουμε οτιδήποτε. Γι' αυτό ε, υπενθυμίζω τους στόχους της ε, χιλιετίας έτσι όπως παρουσιάστηκαν μόνοι τους ε, και όπως αναφέρονται σε αυτή τη μικρή καρτούλα εδώ που κουβαλάω μαζί μου και δείχνω στους ε, ψηφοφόρους είναι πρόκειται για 8 στόχους συγκεκριμένους στόχους πάρα πολύ συγκεκριμένους και πάρα πολύ απλούς θα πρέπει λοιπόν να περιορίσουμε τις φιλοδοξίες μας Λοιπόν, έχω δύο ερωτήσεις να θέσω. Πρώτον, ε, θεμητό εμπόριο, fair trade, πώς μπορούν αυτές οι σχετικές αποφάσεις να συνδυαστούν με τους στόχους της ε, χιλιετίας. Δεύτερη ερώτηση για την πρόσβαση ε, στις ε, στι ναι, διάφορες πηγές ενέργειας ε, ανανεώσιμες ενέργειες ο Μπάνκι Μούν αναφέρθηκε αυτό στην πρόσβαση για όλους σε όλες τις ανανεώσιμες ενέργειες μέχρι το 2030 πως μπορεί να μπει αυτό στους στόχους της χιλιετίας και κάτι τι άλλο να πούμε για τη ε, συνεργασία μας με τις χώρες ΑΚΕ και εν ώψη της μεγάλης συνδιάσκεψης που θα γίνει ε, νομίζω ότι θα πρέπει τα θέματα αυτά που συζητούμε τώρα της, των στόχων της χιλιετίας και τα ε, ε, να τεθούν να συζητηθούν με τις χώρες ΑΚΕ 78 χώρες ΑΚΕ 28 χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό μας δίνει μια τεράστια πλειοψηφία στα Ηνωμένα Έθνη Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι υποφεληθήκαμε από την παρουσία της Επιτρόπου Γεωργίευα ανάμεσά μας και να πω ότι σύμφωνα με τον ΩΣΑ ε, οι φυσικές καταστροφές θα απορροφήσουν ένα πολύ μεγάλο τμήμα του εθνικού ακαθάριστο προϊόντος ε, τα επόμενα χρόνια. Πάντως το θέμα της πρόληψης των φυσικών καταστροφών είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε σοβαρά στις επόμενες συναντήσεις μας και στα πλαίσια των διμερών συζητήσεων που θα έχουμε με άλλες χώρες. Έχει ζητήσει το λόγο ε, επίσης ένα συνάδελφος και μετά θα πάρουν το λόγο οι ομιλητές. Ε, povjerenicima na zaista detaljnom predstavljanju izvješća i politici Europske unije u vezi. Υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα. Υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα και πρέπει να διακόψουμε. Svijetu te mi se čini da je upravo načelo partnerstva sa zemljama koje su najpotrebnije i nema hrvatskog aha je vois que seulement Μόνο ο Επίτροπος Ποτότσνικ κατάφερε να καταλάβει αυτά τα οποία σας είπα στην κροατική γλώσσα. Είναι αλήθεια ότι οι Σλοβαίνοι και οι Κροάτες συνεννοούμεθα μια χαρά και εγώ κατάλαβα πολύ καλά από τον πρωτότυπο τον κύριο Πέτερλε. Θα ήθελα σαν νέο μέλος να ευχαριστήσω τους ε, ε, ε, δύο επιτρόπους για την παρουσίασή τους Πράγματι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος δωρητή στον κόσμο στον τομέα της βοήθειας για την ανάπτυξη και να υπογραμμίσω την αρχή της εταιρική σχέσης με τις χώρες οι οποίες έχουν τις μεγαλύτερε ανάγκες βοήθειας για να πετύχουν τους στόχους του προγράμματος ε, ε, της χιλιετίας των Ηνωμένων Εθνών ε, που δεν έχει πάρα πολλούς πόρους αλλά παρόλα αυτά έχουν καταλάβει ότι πρέπει να κάνουν κάθε προσπάθεια για να επηρεάσουμε τα προγράμματα τα οποία ακολουθούμε ήδη τώρα από το 2005 στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Συνένεσης για την Ανάπτυξη. Θα περάσω τώρα το λόγο στους επιτρόπους Πίμπαλς και Ποτότσνικ, όπως επίσης και στην κυρία Μοχάμετ για να δώσουν τις απαντήσεις τους. Τέσσερα λεπτά ο καθένας. Κύριε Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα αρχίσω με δύο βασικά σημεία. Πιστεύω ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα τα υποστηρίζουμε στεναρά. Είναι και το Ιωβιλέο του I had a dream του Μάρτιν Luther King. Πέρασαν 50 χρόνια. Πριν από 50 χρόνια ήταν αδιανόητο αυτό που είπε και σήμερα είναι εφικτό. Το ίδιο γίνεται και με τα ανθρώπινα ε, δικαιώματα. Πρέπει να πείσουμε τους εταίρους μας ότι αυτό είναι το σωστό. Τι άλλο να κάνουμε, μπορούμε να τους εξαναγκάσουμε, όμως μπορούμε να τους μεταπίσουμε. Και το ίδιο συμβαίνει με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Βλέπουμε στο Νότιο Σουδάν, γενικότερα στην περιοχή της Εχέλ, όλες τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τώρα αρχίζουν να καταλαβαίνουν σιγά σιγά όλοι ότι η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν αποδυναμώνει, ε, ενισχύει, καθιστά ισχυρότερη τη χώρα και ε, είναι βασική παράμετρος ούτως ή άλλως της αναπτυξιακής πολιτικής. Τώρα, σε σχέση με τις επικρίσεις ε, κατά της Ευρώπης, έχω πάει σχεδόν παντού στο, στον κόσμο και δεν υπάρχει καλό και κακό. Ε, απλώς πρέπει να ε, πούμε ότι έχουμε κάνει καλά πράγματα στην Ευρώπη. Κοινωνική ασφάλιση. Ασχολούμαστε με κάθε ανθρώπινη ζωή. Πρέπει λοιπόν όντω να αλλάξουμε, αλλά ας βασιστούμε και στα επιτεύγματά μας. και ε, πιστεύω ότι εκεί στις χώρες και είναι σημαντικό ε, πέρα από τις επικρίσεις ε, να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν υπάρχει ε, σωστό και λάθος, απλώς πάντοτε υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. Αυτή την κατεύθυνση πρέπει να ακολουθήσουμε. Θα ήθελα τώρα να επικεντρωθώ σε κάποια σημεία που ήταν και το αντικείμενο των ερωτήσεών σας. Αυτά που είπε ο Γκέι Μίτσελ και ο κ. Λάστρεμ για τη σημασία ε, της ε, μείωσης ε, των κινδύνων από φυσικές καταστροφές. Μα το σημαντικό είναι να οικοδομήσουμε την ανθεκτικότητα, τη resilience. εντάξει να συμβαζόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τι θα κάνετε, θα φτιάξετε την κυβέρνηση και θα πείτε όχι δεν υλοποιείτε το στόχο αν δεν προστατεύετε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το ίδιο σημαίνει και με τα ενεργειακά προγράμματα. Το βασικό είναι να έχουμε resilience, ανθεκτικότητα, να μπορέσει η χώρα να τα καταφέρει μόνη της και γι' αυτό θα πρέπει να διευρύνουμε την αρχή της μείωσης ε, των κινδύνων των ε, φυσικών καταστροφών. Τώρα, ας περάσω στον κοινό προγραμματισμό. Είναι ζωτική σημασία ε, γιατί έχουμε από 15 και έως 18% των κονδυλίων σε διεθνές επίπεδο και πρέπει να βελτιώσουμε τις επιδόσεις μας, να επιτύχουμε την ευρύτερη δυνατή συνένες των κρατών μελών. Ε, έχουμε 1,8 δις σε ανάληψη υποχρεώσεων στην ε, διάσκεψη της Σομαλίας που ολοκληρώθηκε χτες. Ε, και είναι το καλύτερο που μπορέσαμε να κάνουμε σήμερα, όμως θα ήταν δύσκολο να ισχυριστούμε ότι ότι είναι η πιο αποτελεσματική Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά παρόλα αυτά αυτό πιστεύω αυτή τη στιγμή. Κάποιοι θέλουν να κρατήσουν τους εθνικούς οργανισμούς ε, εν ενεργεία. Εγώ όμως πιστεύω ότι σωστή απάντηση είναι ο κοινό προγραμματισμός. Επειδή δεν έχω και πολύ χρόνο, θα δώσω άλλη μια τελευταία απάντηση για τα δάση. βιώσιμη ανεργία, επιστημιστική ασφάλεια και ενεργειακή ασφάλεια. Αυτά τα τρία σημεία είναι απαραίτητα για να επιβιώσουν τα παρθένα δάση ε, εντάξει, για τη βιοπικιλότητα, τα εθνικά πάρκα και τα λοιπά είναι όλα αυτά πάρα πολύ θετικά, αλλά αυτή είναι βραχυπρόθεσμη στόχη. Εμείς ασχολούμαστε λοιπόν με αυτό και μια πρωτοβουλία που λέγεται FLECT ε, για τη διαχείριση των δασών. Πιστεύω ότι προς το παρόν είναι τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία που έχουν. Περιμένουν περισσότερο από την πρωτοβουλία Red Sin. Αυτά, Πρόεδρε. Εστίασα την προσοχή μου σε κάποια από τα ζητήματα γιατί δεν έχουμε χρόνο για όλα. Ευχαριστώ. Ας ακούσουμε τώρα τον Επίτροπο Ποτόσνικ. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα-πρώτα ε, να απαντήσω κάποιες συγκεκριμένες ερωτήσεις που ετέθησαν με ρώτησε τι κάναμε για να διατηρήσουμε, για να εξασφαλίσουμε βιωσιμότητα. Κοιτάξτε να δείτε, όλες οι πολιτικές που εφαρμόζουμε πάνε προς αυτή την κατεύθυνση. Ό,τι κάναμε στα πλαίσια του Ρίο συν 20 ήταν μέτρα για να εξασφαλίσουν βιωσιμότητα. Ήταν πραγματικά δεν λέω ότι ε, με όλα αυτά που συμφωνήθηκαν συμφωνούσαμε αλλά συνιστούν μια στερεή βάση επί της οποίας μπορούμε να στηριχθούμε για το μέλλον τώρα για το Red Plus και τα σχετικά νομίζω ότι Αυτά είναι καλά παραδείγματα για να δούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα ίδια κονδύλια για διαφορετικές δραστηριότητες, ναι, για, για την κλιματική αλλαγή ή για ε, ακόμη δηλαδή ε, ιδιαίτερα σε μια εποχή κρίσης θα πρέπει να χρησιμοποιούμε τα κονδύλια που έχουμε στη διάθεσή μας για να, αντιμετω, να πετύχουμε άνω του ενός στόχου έτσι για να μπορούμε να κατανείμουμε τα κονδύλια για να επιτύχουμε παραπάνω πράγματα από ένα κοιτάξτε πιστεύω ότι η η βιωσιμότητα δεν περιορίζεται μόνο σε ορισμένους τομείς. Για μένα η βιωσιμότητα είναι ένας γενικότερος όρος που καλύπτει και τα κοινωνικά θέματα και το περιβάλλον κτλ. Ο κύριος Νόιζερ μίλησε για το fair trade. Κοιτάξτε, η παρατήρησή σας κατά την άποψή μου είναι σημαντική γιατί μας καλεί να αρχίσουμε να συζητούμε καινούργια θέματα αλλά θα ήθελα να ξεκαθαρίσω το εξής θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σχετικά με το τι εννοούμε στόχους με την έννοια του goals μακροπρόθεσμους στόχους και βράχοι πρόθεσμους ή μέσο πρόθεσμους στόχους Targets, Goals και targets. Λοιπόν, πώς ορίζουμε αυτά τα δύο πράγματα. Και το από εκεί και πέρα Υπάρχουν πολλά πράγματα για τα οποία ε, πρέπει να, να ε, προσέξουμε ιδιαίτερα. Αυτό που ονομάζουμε στα αγγλικά ownership, δηλαδή το πόσο γίνονται αποδεκτές κάποιες ιδέες, κατά πόσο νεοθετούνται κάποιες απόψεις από τους ενδιαφερόμενους. Όλοι θα οι συμμετέχοντες θα πρέπει να αισθάνονται ότι πράγματι συμμετέχουν και υιοθετούν την όλη φιλοσοφία. Επίσης είναι πολύ σημαντικό Όλε όλες οι οικονομίες είτε σε ανεπτυγμένες χώρες είτε σε αναπτυσσόμενες κτλ. Όλες οι οικονομίες θα πρέπει να υιοθετήσουν την ίδια προσέγγιση για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Όπως είπε και ο κύριος Κατσμάρεκ θα πρέπει να αποφύγουμε λάθη που έγιναν στο παρελθόν και προσθέτω σε αυτό ότι το θεματολόγιο το οποίο περιλαμβάνει θέματα προστασίας του περιβάλλοντος δεν είναι ενάντια στην όλη φιλοσοφία της βιώσιμης ανάπτυξης η, αυτή τη στιγμή η ανάπτυξη που ζούμε στον κόσμο είναι μια ανάπτυξη που έχει συγκεκριμένα όρια εμείς θέλουμε πιο ανοιχτή βιώσιμη ανάπτυξη εν πάση περιπτώσει σας ευχαριστώ όλους σας για την πολύ καλή συζήτηση για την προσέγγιση σας που ε, που θεωρώ εξαιρετική, πολύ καλή. Και τώρα δίνω το λόγο στην κυρία Μινά Μωαμέδη. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη για τις ερωτήσεις και αυτά που είπαν. Εμείς είχαμε κάποιες συγκεκριμένες συνταγές για αυτό που θέλουμε να κάνουμε τώρα, όμως θέλουμε να συζητήσουμε, να επιστρέψουμε στις χώρες μας και να αρχίσουμε να εφαρμόζουμε και να μην ψάχνουμε να βρούμε το τι ακριβώς ε, είχε γίνει και πόσο χρόνο θα χρειαζόμασταν να το εφαρμόσουμε. Το θέμα είναι ότι το πρόγραμμα ήταν πάρα πολύ βαρύ και δεν μπόρεσε να απογειωθεί. Να μην ξεχνάμε οι στόχοι της χιλιετίας ήταν πάρα πολύ χρήσιμοι αλλά παρόλα αυτά σε ορισμένους τομείς είχαμε 150 στόχους. Πώς θα τους επιδιώκαμε όλους αυτούς αν το προσπαθούσαμε. Θα πρέπει λοιπόν να ξεκινήσουμε. Καθορίζοντας καλύτερα τις προτεραιότητές μας, γιατί τα θέματα είναι πάρα πολλά. Η πρόκληση είναι τεράστια. Η συζήτηση η οποία θα πρέπει να ακολουθήσει αφορά 93 χώρες και όλους εμάς εκτός αυτών των χωρών που θα πρέπει να βοηθήσουμε. Να προσπαθήσουμε να βρούμε έναν τρόπο αντιμετώπισης, νέο τρόπο της φτώχειας να αντιμετωπίσουμε τις τεράστιες προκλήσεις και για μας είναι θέμα μετάβασης. Πώς θα βοηθήσουμε να γίνει αυτή η μετάβαση από το σήμερα στο αύριο. Να βοηθήσουμε τους νέους να εμπλακούν γιατί ε, αυτοί θα κουβαλήσουν αυτή την προσπάθεια και θα πρέπει να νιώσουν ότι είναι δική τους αυτή η προσπάθεια. Έτσι λοιπόν τα κομβικά σημεία με τα οποία θα μετακινηθούμε θα βοηθήσουν να πετύχουμε τους στόχους. Έχουμε κάνει προσπάθεια, ε, αλλά παρόλα αυτά πολλά μένει να γίνουν. Νομίζω ότι έχουμε αρχίσει αυτή τη στιγμή να σχεδιάζουμε το περίγραμμα ε, των προσπαθειών μας. Δεν πρέπει να εγκαταλείψουμε κανέναν πίσω, δεν πρέπει να καθυστερήσουμε κανέναν και δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να ιεραρχήσουμε τα δικαιώματα των ανθρώπων αυτής της γης, γιατί εδώ η ισότητα όλων είναι δεδομένη. Πρέπει λοιπόν να κρατήσουμε τον στόχο, τη μηδενική πείνα, τα δικαιώματα και των ε, ομοφιλόφιλων ανδρών και γυναικών κλπ. Η προσπάθεια αυτή έχει πετύχει σε ορισμένες χώρες περισσότερο από ό,τι σε άλλες. Αλλά παρόλα αυτά και η ειδική εκπρόσωπός μας, η κυρία Βάλστρομ, έχει μπορέσει να προχωρήσει ε, στην καταγραφή κάποιων επιτυχιών που με τη σειρά τους θα βοηθήσουν να καθορίσουμε καλύτερα τη στρατηγική μας στο μέλλον. Υπάρχουν λοιπόν προσπάθειες που μένει να γίνουν, θέματα όπως η ενέργεια για όλους, οι συνέπειες των κλιματολογικών αλλαγών, είναι, σαφή ότι, είναι σαφές ότι πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε και θέματα εμπορικά και θα πρέπει όλα αυτά τα θέματα να μην είναι μόνο θέματα συζήτησης αλλά και να περάσουμε σε εφαρμογές των αποφάσεων. Να πω επίσης ότι είχαμε μια τεράστια ευκαιρία στη χώρα μου στην Ιγυρία όπου δεν, παίξαμε, δεν δώσαμε ποτέ ιδιαίτερο βάρος στο θέμα του περιβάλλοντος. Αλλά όταν επισκεφθήκαμε εμείς αυτό το πρόγραμμα είδαμε ότι μας άνοιξε νέες προοπτικές για το τι μπορούσαμε να κάνουμε σε άλλες περιοχές της χώρας, για το περιβάλλον, την οικονομία και κυρίως τους ανθρώπους. Είναι λοιπόν μια άξια πρωτοβουλία, είναι ένα παράδειγμα πρωτοβουλίας που πέτυχε και πρέπει να μιμηθούμε. Ευχαριστώ. Προτείνω στον κύριο Γκρότε τώρα την τελική του παρέμβαση. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι για μένα τουλάχιστον προσωπικά ήταν ένα απόγευμα που μου έμαθε πολλά πράγματα άκουσα αυτά που ελέγχθησαν ότι θα πρέπει όπως είπε και η κυρία Μοχάμεν, ότι θα πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι να είμαστε συγκεκριμένοι στο πώς θα υλοποιήσουμε τους στόχους και συγκεκριμένοι όσον αφορά τη χρηματοδότηση να υπάρχουν σαφείς ε, οδηγίες σαφείς δηλώσεις σχετικά με το τι θα γίνει από αυτά που είπαν οι Επιτρόποι κατέστη σαφές δεν κάθονται βέβαια δίπλα ο ένας με τον άλλον και δεν είδα να περνάει κανένα χαρτί από τον έναν στον άλλον αλλά είναι προφανές ποια είναι η θέση ολόκληρης της Κομισιόν αν θέλετε ή και των δύο ε, επιτρόπων και πραγματικά θα πρέπει ε, όλοι μας να ε, προσπαθήσουμε να απλουστεύσουμε τα πράγματα του ώστε να μας καταλάβει και ο κόσμος ε, η κάρτα που έδειξε ο Νόιζερ ήταν ένα καλό παράδειγμα νομίζω ε, πάντως για μένα δεν είναι μόνο ο, η Επιτροπή Περιβάλλοντος είναι και η Επιτροπή ε, Υγείας για και άλλες επιτροπές που μπορούν να συμμετάσχουν σε μια κοινή προσπάθεια για να ξεκινήσουμε τη συζήτηση για ορισμένα θέματα. Παραδείγματο χάρη βιοκαύσιμα. Αν προωθηθούν τα βιοκαύσιμα, ε, πώς, αυτό πώς επηρεάζει τα πράγματα σε άλλες περιοχές του κόσμου. Αν ε, πετάμε το 50% των τροφίμων μας ε, αυτό πώς επηρεάζει τον υπόλοιπο κόσμο αυτά για τα δάση ένα άλλο τεράστιο θέμα Επίσης η εμπορική πολιτική αναφέρθηκε επανειλημμένα σήμερα η εμπορική πολιτική φτιάχνει μια γέφυρα προς τη βιωσιμότητα. Η συνθήκη της Λισαβόνας μας δίνει τη δυνατότητα να συμφωνήσουμε ή να απορρίψουμε ορισμένα πράγματα και ε, νομίζω ότι έχουμε τη δυνατότητα να ε, υλοποιήσουμε στόχους για να προωθήσουμε αν θέλετε μια βιωσιμότητα και σε άλλες περιοχές του κόσμου. Σας ευχαριστώ πολύ για όλα αυτά που μου μάθατε σήμερα, ιδιαίτερα την κυρία Μοχάμεν, τον κύριο Ποτότσνικ, τον κύριο Πίμπαλξ και όλους εσάς και όλα τα μέλη της Επιτροπής για την κοινή αυτή συνάντηση. Είναι μια αρχή νομίζω. Πρόεδρος, και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω από πλευρά μου την κυρία Μωαμέτ, τον κύριο Γκρότε, την ε, Επιτροπή Περιβάλλοντος και τα, τον κύριο Πίπαλ και τον κύριο Πουτότσινγκ που βρίσκονταν εδώ για να συζητήσουμε μαζί μας ένα τόσο σοβαρό θέμα. Όπως θα τονίσει και ο κύριος Μπάνκι Μουν στην επόμενη σύνοδο των Ηνωμένων Εθνών, χρειαζόμαστε μια καινούρια προσέγγιση θέλουμε να προωθήσουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη την οποία θα και θα πρέπει να δουλέψουμε με ένα καινούριο τρόπο. Αυτό σημαίνει δουλειά από πλευρά όλων μας, καινούριες προσπάθειες αλλά καινούργια συνεργασία σε πλανητικό επίπεδο. Ευχαριστώ πολύ. Je Σας υπενθυμίζω δεν ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση. Αποχωρήστε σας παρακαλώ με ησυχία γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί η συνεδρίαση όπως έλεγα.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 για το προσχέδιο νομοδότησης για την Επιτροπή Προϋπολογισμών για το 2014. Σας θυμίζω ότι κατά τη διάρκεια της συναδριώσεων μας στις 28 Αυγούστου υιοθετήσαμε τις τροπολογίες μας και τώρα θα πρέπει να συζητήσουμε το θέμα της νομοδότησης που αναφέρεται σε μια έκθεση την οποία προετοιμάζει η Επιτροπή Προϋπολογισμών. Θα ψηφιστεί στις 9 Οκτωβρίου η έκθεση αυτή. Η δημοσιονομική διαδικασία φέτος άργησε και δεν έχουμε ακόμα καταφέρει να ανακτήσουμε την καθυστέρηση αυτή. Έχουμε το σχέδιο μόνο στα αγγλικά. Η συγητής μας είναι ο Ρικάρντο Κορτές Λάστρα και του δίνω το λόγο. <coughs> Κύριε Κορτές Λάστρα, έχετε το λόγο. Ε, τέσσερις βασικές γραμμές για να παρουσιάσω αυτή τη γνωμοδότηση η οποία νομίζω ανταποκρίνεται με τις θέσεις τις οποίες ήδη είχε η Επιτροπή μας στις 28 Αυγούστου όταν ψηφίσαμε τις βασικές τροπολογίες για το 2014, για τον προϋπολογισμό του 2014. Ε, στην ουσία θέλουμε περισσότερους πόρους για την ανάπτυξη. Αυτό είναι ο βασικός στόχος. Εμείς επιμένουμε λοιπόν στην ανάγκη η οποία υπάρχει να μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους τους οποίους έχουμε θέσει σαν Επιτροπή Ανάπτυξη. Από την άλλη τους στόχους της χιλιετίας, όλο αυτό συζητούσαμε σήμερα, και από την άλλη θέλουμε να αυξήσουμε το εσωτερικό ακαθάριστο προϊόν. Δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να θυγούν ακόμα περισσότερο αυτοί οι οποίοι ήδη υποφέρουν από την κρίση η οποία σοβεί. Θα πρέπει λοιπόν εδώ να προσπαθήσουμε να στηρίξουμε μία πρόταση προϋπολογισμού αντίστοιχου τουλάχιστον με το 2013. Πέραν αυτού αυτό το οποίο θέλουμε είναι να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια στην εκτέλεση του προϋπολογισμού αυτού. Θέλουμε να διατηρηθούν οι γραμμές του προϋπολογισμού όσοι είχαν. Σήμερα το πρωί είχαμε μία συνάντηση με την εισηγήτρια της Επιτροπής Προϋπολογισμών και ε, συμφωνεί και αυτή ότι θα προσπαθήσει να κρατήσει τα επίπεδα τις γραμμές αυτές τα επίπεδα τα οποία είχαν τον προηγούμενο χρόνο. Εδώ θα υπάρξει υποστήριξη από όλες τις πολιτικές ομάδες. Τελικά να υπάρξουν περισσότεροι πόροι για την ανάπτυξη και τη συνεργασία. Πολύ σας ευχαριστούμε κύριε Κόρτες Λάστρα. Δεν ζητάει κανείς το λόγο. Ας ακούσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Si elle le souhaite. Αν θέλετε βεβαίως. Ε, κοιτάξτε, ήθελα μόνο να ευχαριστήσω εξ ονόμας Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, την Επιτροπή Ανάπτυξης ε, για όλη τη δουλειά που έχουν κάνει για τον προϋπολογισμό. Όπως ξέρετε, είναι προϋπολογισμός κρίσης. Και περιεκόπησε σε σημαντικό βαθμό κατά την εξέταση του Συμβουλίου. Όπως είπε και ο εισηγητής, ο στόχος ε, του προϋπολογισμού είναι η εκπλήρωση των βασικών ε, στόχων ε, για τα απτυξιακά ζητήματα για τα οποία συζητήσαμε επί μακρόν στην προηγούμενη ακρόαση και ε, στοχεύει επίσης τους πλέον άπορους της Ένωσης. Αναθεωρήθηκε άρδιν ε, ο προϋπολογισμός ως προς την ε, δημοσιονομική ονοματολογία για δύο λόγους. Πρώτον, για να επιδείχουμε μεγαλύτερη διαφάνεια. Ορισμένες φορές δεν γίνεται κατανοητό ότι Συντάξαμε αυτό το προπολογισμό για να ε, βλέπουμε καλύτερα τα αποτελέσματα, να μετρούμε τις επιδόσεις και σε κάθε γραμμή του προϋπολογισμού έχουμε δείκτες ε, επιδόσεις, επιδόσεων. Και ε, επιδιώκουμε μεγαλύτερη ευελιξία και βελτιστοποίηση της χρήσης των κονδυλίων. Είναι τον όνου κάνευ σήμερα η ευελιξία αυτή. Εάν ε, προκύψει κάποια κρίση είναι εύκολο να μεταφέρονται επιστώσεις από τη μία γραμμή στην άλλη και ε, σε περίπτωση απρόβλεπτων δράσεων πρέπει όμως να αναλυφθούν. Μπορούμε σε εισαγωγικά να παίξουμε με τις γραμμές του προϋπολογισμού, τόσο ώστε να έχουμε βελτιστοποιημένη απορρόφηση και χρήση των κονδυλίων. Κύριε Κορτιζλάς, θα θέλετε το λόγο, ρωτάει η Πρόεδρος. Όχι, λοιπόν. Για το σχέδιο έχουμε καταληκτική ημερομηνία 18 Σεπτεμβρίου, 12 το μεσημέρι. Τελευταίο σημείο ουσιαστικό της ημερήσιας διάταξης ε, Έχουμε ανταλλαγή απόψεων με εκπροσώπους των τεσσάρων βασικότερων περιφερειακών οργανώσεων της Ανατολικής Αφρικής. Ήρθαν για τη διάσκεψη για τη Σομαλία που έλαβε χώρα εχθές, αλλά ήρθαν και σε εμά για ανταλλαγή απόψεων. Η ανταλλαγή απόψεων εγγράφεται στο πλαίσιο του ενδιαφέροντος που έχει η Επιτροπή μας για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης που υποστηρίζει την περιφερειακή ολοκλήρωση μεταξύ άλλων στην Αφρική. Ε, έχουμε την κοινότητα Ανατολικής ε, και μεσημβρινής Αφρικής ε, και στα πλαίσια της Συμφωνίας ε, του Κοτονού έχουμε το πλαίσιο συνεργασίας ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις τέσσερις περιφερειακές οργανώσεις η κοινότητα της Ανατολικής Αφρικής, η Διακυβερνητική Αρχή για την Ανάπτυξη, η Επιτροπή του Ινδικού Ωκεανού και η κοινή αγορά της Ανατολικής και Μεσημβρινής Αφρικής. Αρχικά 619 εκατομμύρια έχουν προβλεφθεί για δύο βασικούς τομείς. Πρώτον, οικονομική, περιφερειακή οικονομική ολοκλήρωση και δεύτερος στόχος, πολιτική περιφερειακή ολοκλήρωση. Όμως, 193 εκατομμύρια από αυτά τα αρχικά κονδύλια πέρυσι διοχετεύτηκαν στην πρωτοβουλία ε, βιώσιμη ενέργεια για όλους. Ε, ξέρετε ότι τώρα γίνεται η ενδέκατη αναθεώρηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης ε, θα θέλαμε να ακούσουμε από του εκπροσώπου αυτών των οργανώσεων αν επωφελήθηκαν από αυτή την υποστήριξη και ποια είναι κατά τη γνώμη του τα προσκόμματα που θα υπήρχαν και που εμποδίζουν την πολιτική και οικονομική περιφερειακή ολοκλήρωση στην Ανατολική Αφρική. Ζητώ συγγνώμη να παραφθείρω κάποια ονόματα. Καλωσορίζω τον κύριο Γουένια, που είναι Γενικό Γραμματέα ε, ε, τη Κοινή Αγορά Ανατολική και Μεσηβρινή ε, Αφρική, ο κύριο Ρίτσαρτ Ζεζίμπερα, Γενικό Γραμματέα Κοινότητα Ανατολική Αφρική, ο κύριο Μαχμούντ Μαλίμ, εκτελεστικό γραμματέα της Διακυβερνητική Αρχής για την Ανάπτυξη και τέλος ο κύριος Ζαν Κλοντ Λεστχάκ, Γενικός Γραμματέας Επιτροπής του Ινδικού Ωκεανού Εξοχότατε Ρίτσαρντ ε, Σέτσι Μπεράι, ε, ε, τελείται καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της Κοινότητας Ανατολικής Αφρικής. Έχετε πρώτος το λόγο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και εσάς και τα, ε, τους άλλους ευρωβουλευτές που είναι μέλη της Επιτροπής Ανάπτυξης, που είναι μέλη της των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, θα ήθελα να κάνω ε, εδώ μια δήλωση εκ μέρους και των συναδέλφων από άλλες επιτροπές από την Επιτροπή του Ειδικού Οκεανού, από την Ίγκατα, από την Κομέσα η περιοχή, η περιοχή μας καλύπτει ουσιαστικά το πάνω από το 50% του πληθυσμού της Αφρικής πάνω από το ίμιση του εδάφους και περιλαμβάνει και την, τις περιοχές με τη μεγαλύτερη ανάπτυξη όχι μόνο στην Αφρικανική Ήπειρο αλλά στον κόσμο ολόκληρο. Έξι από τις ε, γρηγορότερα αναπτυσσόμενες χώρες στον κόσμο βρίσκονται στην περιοχή μας και η περιοχή μας έζησε εδώ και δεκαετίες κάθε χρόνο ε, εμβάθυνση της ε, συνεργασίας και της ξέρουμε βεβαίως ότι η Ευρώπη υποστηρίζει αυτή την όλο και στενότερη σχέση μεταξύ των χωρών ΑΚΕ και της Υπήρου μας και αλλού η περιφερειακή συνεργασία και η περιφερειακή ενσωμάτωση είναι βασική στόχη και για την Ευρώπη εκποφεληθήκαμε από το EDF 9, από το EDF 10 και τώρα βρισκόμαστε στο EDF 11 το Ταμείο Ανάπτυξης το Ευρωπαϊκό Ταμείο με συγχωρείτε Ανάπτυξης το ΦΕΝΤΕΡ αλλά προσπαθούμε και εμείς να ενισχύσουμε την ανάπτυξή μας προσπαθούμε και εμείς να κάνουμε προσπάθειες και να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό η σημαντική πάντα η συνεργασία με την Ευρώπη η οποία αποδίδει καρπούς και για την Αφρική αλλά και για την Ευρώπη μέσα στα πλαίσια του EDF 10 είχαμε την ευκαιρία να επενδύσουμε στη σε, θέματα ειρήνης και ασφάλειας φυσικών ε, ε, πόρων και κρίσιμων υποδομών. Ο συνάδελφος από την ΕΓΚΑΤ ήταν εδώ τις τελευταίες δύο μέρες ε, και συζήτησε τα θέματα της Σομαλίας. Η περιοχή μας έπαιξε σημαντικό ρόλο για την ενίσχυση της ειρήνης και της ασφάλειας όχι μόνο στη Σομαλία αλλά και για την ενίσχυση της και ε, της ασφάλειας στον Ινδικό ωκεανό και ε, προωθήθηκαν προγράμματα με σημαντική στήριξη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσον αφορά τώρα τους φυσικούς πόρους, με μεγάλη χαρά σας λέω ότι η Ινδική Επιτροπή με στήριξη Ευρωπαϊκής Ένωσης κατάφερε να συνεισφέρει στην ανάπτυξη ε, πολλών οικογενειών, πάνω από 3,5 εκατομμύρια ήταν αυτές οι οικογένειες, μάλλον να κατάφερε να συνεισφέρει στην ασφάλεια των τροφίμων αυτών των οικογενειών. Ξέρουμε πολύ καλά ότι τέτοιου είδους στήριξη και βοήθεια βοηθάει ολόκληρη την περιοχή και η υποστήριξη τον αγώνα κατά της πειρατείας στη θάλασσα είναι επίσης πολύ σημαντική και έτσι μπορέσαμε να αναπτύξουμε ε, να αναπτύξουμε και 5 εκατομμύρια ε, τετραγωνικά χιλιόμετρα του Ινδικού ωκεανού αυτού καθεαυτού. Εμείς υποστηρίζουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επενδύουμε και προσπαθούμε να ενισχύσουμε την δηλωνιακή μας ένωση προσπαθούμε να φτιάξουμε μια ενιαία εσωτερική αγορά και καταφέραμε να κάνουμε σημαντική πρόοδο σχετικά με μια νομισματική ένωση θα ήθελα επίσης να σας πω ότι για τις υποδομές και για τις ανανεώσιμες ενέργειες με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα πλαίσια του EDF 10 έγιναν μεγάλες πρόοδοι στον ενεργειακό τομέα, στο τομέα των οδών και αυτοκινητοδρόμων και στον τομέα του εμπορίου. Και τέλος, αυτή η στρατηγική εταιρική σχέση με την Ευρώπη δεν ε, είναι ξεκομμένη από τις δικές μας προσπάθειες. Η ΣΑΝΤΕΚ, η ΚΟΜΕΣΑ συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις για τη δημιουργία μιας τριμερούς εμπορικής ένωσης που ελπίζουμε να ευοδοθεί. Επίσης και στο ΕΓΚΑΤ και στην τριμερή ασχολούμεθα και με προγράμματα υποδομών και μεταφορών τα οποία πιστεύουμε ότι θα μπορέσουν να ξεκλειδώσουν το πλήρες δυναμικό της περιοχής μας. Και τέλος η συνεργασία μας είναι βασισμένη στην ανάγκη ε, ανάπτυξης καλής διακυβέρνησης, δημοκρατίας και ασφάλειας στην περιοχή. Πραγματικά περιμένω με ανυπομονησία τις συζητήσεις που θα γίνουν για το EDF 11 και θα θέλαμε ακόμη μια πιο στενή και βαθιά συνεργασία μεταξύ της περιοχής μας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν έχει ζητήσει το λόγο κάποιος συνάδελφος. Όχι. Από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχετε το λόγο. Ευχαριστούμε, Πρόεδρε. Εκπροσωπώ, προς μεγάλη μου χαρά, την, την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και ταυτόχρονα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η ασφάλεια, η σταθερότητα, η ασφάλεια και η διακυβέρνηση στην Αφρική ε, είναι βασικό μέλημα και της Επιτροπής και της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης γιατί πρόκειται για στρατηγικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εξασφάλιση της σταθερότητα και της ασφάλειας θα επιτρέψει κοινωνικονομική ανάπτυξη για την καταπολέμηση της στόχης και την αύξηση του επίπεδου διαβίωσης. Επίσης θα τονώσει την περιφερειακή, οικονομική, κοινωνική και πολιτική ολοκλήρωση και θα δημιουργήσει και περιφερειακή νέα δυναμική ε, για την ε, αντιμετώπιση των ενόπλων σειράξεων. Λοιπόν, ε, για την ε, τόνωση της ασφάλειας ε, και της σταθερότητας αντιλαμβανόμαστε ότι ο πολιτικός διάλογος δεν μπορεί να προχωρήσει ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους Αφρικανούς εταίρους της αν δεν εξασφαλιστεί η ασφάλεια και η σταθερότητα κατά προτεραιότητα. Το ίδιο ισχύει φυσικά για την περιοχή του Ινδικού και του Ειρηνικού. Οι περιφερειακές οργανώσεις είναι ήδη πολύ σημαντικός πυλώνας της αρχιτεκτονικής ασφάλειας και ε, σταθερότητας ε, της Αφρικής που υποστηρίζεται από το Africa Peace Facility ή από την Αφρικανική Ένωση. Στο κέρας της Αφρικής, παραδείγματος χάρη, εμπλέκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι έχει υιοθετήσει στρατηγικό πλαίσιο για το κέρας της Αφρικής. Έχει διορίσει ακόμη και ειδικό εκπρόσωπο ε, για αυτήν την περιοχή στο κέρας ε, της Αφρικής. Έχουμε μια σφαιρική και ολοκληρωμένη προσέγγιση με διασυνδεδεμένα όλα τα διαθέσιμα εργαλεία, είτε είναι πολιτικά ή σχετίζονται με την ασφάλεια ή το εμπόριο. Στη διάσκεψη για τη Σομαλία, όπου συμπροέδρευσε η ύπατη εκπρόσωπος και ο πρόεδρος της Σομαλίας, Είδαμε αυτές αποδείξεις της ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής προσέγγισης θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε άοκνα για να επιτύχουμε περιφερειακή ολοκλήρωση στην Αφρική και με τη βοήθεια της ΙΚΑΤ φυσικά. Ποιες είναι οι προσδοκίες μας για τις περιφερειακές οργανώσεις. First, the EU's relationship with the African σχέση με την υποσαχάρια Αφρική. Πρέπει να διέπονται από μια στρατηγική πολιτική θεώρηση των πραγμάτων και να βασιζόμαστε σε μια ρεαλιστική στρατηγική περιφερειακής ολοκλήρωσης όπου οι περιφερειακές οργανώσεις και τα μέλη τους θα έχουν αναλάβει εξίσου δέσμευση. Χωρίς αυτές τις απτές δεσμεύσεις σε εθνικό επίπεδο πιστεύουμε ότι η περιφερειακή ολοκλήρωση δεν είναι υλοποιήσιμη. Δεύτερον, οι περιφερειακές οργανώσεις πρέπει να είναι ζωντανές ε, και ναι, δραστήριες ε, για να εκπληρώσουν τους στόχους σα. Ε, και χρειάζεται απόλυτη δέσμευση από πλευρά των κρατών μελών για την επίτευξη των στόχων με την 11η αναθεώρηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης και σε συνεργασία με τις περιφερειακές οργανώσεις στην περιοχή του Ειρηνικού είτε του Ατλαντικού και για πολλά θέματα μεταξύ των οποίων και ανάπτυξη ενδογενών ικανοτήτων. Ε, χρειαζόμαστε καλή επικοινωνιακή πολιτική επίσης στη σχέση μας με τις περιφερειακές οργανώσεις ε, και υπάρχει ειδική εντολή για αυτό. Έχω και δύο συναδέλφους ε, εδώ που εργάζονται σε περιφερειακές ε, επιτόπου, δηλαδή αντιπροσωπείες Ευρωπαϊκής Ένωσης, τακτικές συναντήσεις σε υπουργικό επίπεδο με τις περιφερειακές οργανώσεις εμβαθύνει τον πολιτικό διάλογο για την περιφερειακή πολιτικο-οικονομική ολοκλήρωση και τέλος προτείναμε μια νέα προσέγγιση για τον ε, προγραμματισμό των ε, υποταμείων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξη. Αρχίσαμε ένα νέο διάλογο με του εταίρου μα για αυτή τη νέα προσέγγιση και είμαστε πεπισμένοι ότι θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε για τους καλύτερους όρους ε, εφαρμογής του 10 ου ενδεικτικού περιφερειακού προγράμματος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης. Πολύ σας ευχαριστούμε. Η κυρία Σαγεντίνη έχει ζητήσει το λόγο. Σας ακούμε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, είχα την εντύπωση εγώ ότι θα ακούγαμε όλους τους. Και ίσως βέβαια και αυτά που θα πω τώρα να τα λάβουν υπόψη οι επόμενοι ε, ομιλητές. Μπορούμε να είμαστε ευγενείς μεταξύ μας και να μας πείτε ότι η συνεργασία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις χώρες της ε, ε, νότιο-ανατολικής Αφρικής πάνε μια χαρά και για τη νέα περίοδο του EDF. Αλλά σήμερα το πρωί είχαμε μια ακρόαση σε αυτό το κοινοβούλιο σχετικά με την διαφάνεια σε θέματα σαν παράδειγμα πρώτων υλών και όπως είπα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει θα έλεγα συνεκτικότητα στους στόχους μας έτσι ώστε όλες οι πολιτικές να μην ε, ε, είναι επιβλαβής για την αναπτυξιακή πολιτική, ίσα ίσα να την βελτιώνουν. Θα ήθελα λοιπόν να μας πείτε με κάθε ειλικρίνεια τη συνεργασία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ανατολική Αφρική, όχι μόνο πάνω στα θέματα ε, που αφορούν το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης. Εμείς σαν Κοινοβουλευτική Επιτροπή είχαμε καταψηφίσει ε, την πολιτική ε, για την Ανατολική Αφρική μετά από δική μου πρόταση, ήμουν εισηγήτρια τότε. Αυτό είναι κάτι το οποίο όμως δεν έγινε ε, δεκτό σαν πρόταση από τους συναδέλφους της Επιτροπής Διεθνού Εμπορίου. Αλλά εμεί θεωρήσαμε ότι το EPA για την Ανατολική Αφρική δεν ήταν σωστό και δεν καθιέρωνε αυτό που θα θέλαμε εμείς να είναι μια πραγματική εταιρική σχέση αλλά ήταν μια απλή εμπορική συμφωνία. Πιστεύω εμείς ότι από τέτοιους ε, ε, ανταλλαγές απόψεων μπορούμε όλοι να κερδίσουμε, εφόσον μας πείτε πώς πάνε τα πράγματα επί τόπου, πώς ε, οι συμφωνίες αυτές, οι συμφωνίες οι επενδυτικές, σαν παράδειγμα, πώς θα έλεγα λειτουργούν επί στην Ανατολική Αφρική και πώς μπορούμε εμείς να διασφαλίσουμε τη συνεκτικότητα των πολιτικών μας. Θα αναφερθώ σε ένα θέμα ανεκδοτολογικά που δεν αφορά την Ανατολική Αφρική. Είχα ασχοληθεί και με την αντίστοιχη συμφωνία για την ε, Κεντρική Αφρική και όταν είχε προχωρήσει η συζήτηση στην Επιτροπή Εμπορίου, Διεθνούς Εμπορίου μάλλον, ο πρέσβης του Καμερούν ήταν παρόν και δεν είπε τίποτα. Δεν είπε αυτό το οποίο θα έλεγε αργότερα ότι δεν είναι καθόλου ε, ε, ικανοποιημένοι από την ενδιάμεση συμφωνία. Άμα δεν μας πείτε ακριβώς, ε, δεν μπορούμε εμείς να το μαντέψουμε, δεν θέλουμε να είμαστε πατερναλιστές, θέλουμε να κάνουμε αυτό το οποίο και εσείς θέλετε. Τα προγράμματα αυτά είναι ιδιαίτερα πατερναλιστικά για την κεντρική Αφρική. Μπορεί να θυμώσετε μαζί μου γιατί το διαπίστωσα και εγώ αυτό, αλλά νομίζω ότι έτσι πρέπει να είναι οι συζητήσεις ειλικρινείς μεταξύ μας και ελπίζω ότι οι επόμενοι ομιλητές να είναι και αυτοί απόλυτα ειλικρινείς και ίσως να μας πούνε κάπως περισσότερα από αυτά τα οποία εσείς μας είπατε. Δεν ξέρω, θέλετε όλοι να απαντήσετε. Ποιος θέλει να πάει πρώτος στο λόγο. Ευχαριστώ. να ασχοληθώ με δύο θέματα πάρα πολύ σύντομα με πάρα πολύ απλοϊκό και ε, θα έλεγα ειλικρινή τρόπο. Ξέρουμε που είναι τα προβλήματα. That uh, within the context of the interim uh, EPAs, uh, you have the EU raw material initiative. Σχετικά με τις συμφωνίες εμπορικές για τα βασικά προϊόντα, ε, για την ε, μη επιβολή περαιτέρω φορολογικών επιβαρύνσεων στις εξαγωγές. Όλοι γνωρίζουμε ότι ε, υπάρχουν οι φόροι αυτοί για αναπτυξιακούς λόγους. Είναι θέμα το οποίο θα έλεγα είναι κατά προτεραιότητα αντιμετωπίσιμο και εμείς είμαστε ευχαριστημένοι γιατί κάποιοι από εμά ήδη από το 70 είχαμε σημειώσει το πρόβλημα και είδαμε κάποιες επιχειρήσεις διεθνείς όπως η Amazon τι κάνει για να αποφεύγει να πληρώνει ευρωπαϊκούς φόρους, ίσως να κατανοήσουν οι Ευρωπαίοι πώς ε, έχει η κατάσταση. Πάντως μπορώ να σας πω εδώ ότι η πλειοψηφία των χωρών θεωρεί ότι οι συμφωνίες αυτές είναι μερκαντιλιστικού τύπου, όχι απλά ελευθέρου εμπορίου, όπου ο μεγάλος εταίρος είναι αυτός ο οποίος απλά επιβάλλει τους όρους του, δεν είναι αναπτυξιακή η συμφωνία αυτή. Με τα δεν έχουμε ε, κάποια προβλήματα. Εμείς ε, πιστεύουμε ότι λειτουργούν αναπτυξιακά. Αλλά αυτό το οποίο μπορώ να σας πω σε σχέση με την αδυναμία της ευρωπαϊκής τάσης είναι ότι η Ευρώπη έχει μια παλιά σχέση με τις χώρες ΑΚΕ, με τις χώρες ιδιαίτερα της Ανατολικής και Νότιας Αφρικής και μερικές φορές εμείς τις προσπάθειες και συμφωνίες που έχουμε υπογράψει δεν έχουμε εντάξει τον ιδιωτικό τομέα. Όταν βλέπω πως η Ιαπωνία σαν παράδειγμα προχωρά σε συμφωνίες και σε εταιρικές σχέσεις προβλέπει τον ιδιωτικό τομέα. Ξέρω ότι χρειάζεται ε, να δραστηριοποιηθεί και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έτσι ώστε και ο ευρωπαϊκός ιδιωτικός τομέας να συμμετέχει περισσότερο. Είναι μια αδυναμία εδώ και εγώ την ερμηνεύω από το ότι η προσπάθεια που γίνεται είναι γραφειοκρατική και δεν είναι εύκολα επηρεάσιμη έτσι ώστε να είναι παρόν ο ιδιωτικός τομέας και στην Ευρώπη και στις περιοχές της Αφρικής προς όφελος όλων. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελε κάποιος να προσθέσει κάτι. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η σχέση ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε εμά είναι καλές και εγκάρδιες και μάλιστα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να πούμε όμως εδώ ότι και στις καλές σχέσεις πάντα υπάρχει χώρος βελτίωσης. Εκτιμούμε το ότι εσείς γενναιόδωρα εγκρίνατε το νέο πακέτο για το νέο αναπτυξιακό κύκλο, ο οποίος τώρα μπαίνει στην αρχική διαδικασία. Έχετε και εσείς τα δικά σας προβλήματα, έχετε θέματα λιτότητας και στις δικές σας χώρες. Είναι κάτι το οποίο έχει ήδη αναφερθεί. Εμείς ε, έχουμε ξεκινήσει τις συναντήσεις μας, είχαμε συναντήσεις και νωρίτερα και μέχρι το τέλος της εβδομάδας και θέλουμε να καλυφθεί πλήρως, ε, να υπάρξει μια πλήρη συμφωνία για την κάλυψη των αναγκών του νέου αναπτυξιακού κύκλου και προσπαθούμε να εμπλουτίσουμε τη διαδικασία αυτή και πώς είναι εφαρμόσιμες οι κατευθυντήριες γραμμές και πώς μπορούμε να συνδυάσουμε τις προσπάθειες αυτές. Χαίρομαι λοιπόν που έχουμε αυτή τη δυνατότητα και χαίρομαι που η συνάδελφος να, προσπαθεί να προκαλέσει μια ουσιαστικότερη συζήτηση. Πάντως, στα πλαίσια της αρχιτεκτονικής ειρήνης και ασφάλειας, αυτό είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό και για τη δική μας περιοχή. Είναι μια περιοχή στην οποία εμπλέκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και πάρα πολύ καιρό. Η χρηματοδότηση πρέπει να στηρίξει προσπάθειες όπως σαν παράδειγμα η εκπαίδευση των ενόπλων δυνάμεων και των δυνάμεων ασφαλείας στην Σομαλία. και να προχωρήσουμε σε χρηματοδότηση ενεργειών και στον τομέα της πρόληψης συγκρούσεων, ε, δίωξης ε, των εγκληματικών ενεργειών, δημιουργίας μέσων ε, μέτρων για την ανάπτυξη της αμοιβαίας εμπιστοσύνης Just one Αναφερθήκατε και για την ενδιάμεση ΕΠΑ, e την ενδιάμεση συμφωνία. Να ήθελα να πω ότι ότι θα διαπραγματευτούμε ε, μια τέτοια συμφωνία για τα επόμενα τρία χρόνια. Έχουμε ένα σύστημα το οποίο θα πρέπει να λειτουργήσει και σε επίπεδο αναπτυξιακής στρατηγικής και θα ενισχύει την περιφερειακή ολοκλήρωση και ταυτόχρονα έχουμε προσπαθήσει έτσι ώστε σε αυτά τα θέματα όταν η Αφρική θα πρέπει να προστατεύεται θα πρέπει να τα φέρνουμε στην επιφάνεια. Γι' αυτό και δεν έχουμε κλείσει το θέμα αυτό. Έχουμε πολλά να κάνουμε και σε επίπεδο MFM και σε επίπεδο ε, τελωνιακών δασμών. Θέλουμε επίσης ε, να μην μας επιβάλλει με το ζόρι πράγματα η Ευρώπη. Θέλουμε να υπάρξει σωστή διαπραγμάτευση των εμπορικών σχέσεων ανάμεσα στην Ανατολική Αφρική και την Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ε, δίστασα να πάρω το λόγο, γιατί η Επιτροπή του Ινδικού ξέρετε ότι είναι μια ομάδα, η μοναδική ομάδα μάλλον, νήσων, ...την Αφρικανική περιοχή, περιφέρεια γενικότερα. Και γι' αυτό αντιμετωπίζουμε κάποια προβλήματα σχετικά διαφορετικά από τα αντίστοιχα της υπηρετικής ε, περιοχής, δηλαδή της υπόλοιπης Αφρικής. Και γι' αυτό αυτά τα οποία μπορώ να σας πω ίσως ε, να ε, θεωρηθούν σαν μια διαφορά ανάμεσά μας. Δεν ισχύει αυτό. Απλά έχουμε κάποια θέματα, κάποια προβλήματα πολύ διαφορετικά τα οποία δεν αντιμετωπίζουν οι χώρες της Υπηρετικής Αφρικής. Και γι' αυτό ακριβώς στον τομέα της ανάπτυξης ακολουθούμε μία στρατηγική η οποία είναι διαφορετική από την αντίστοιχη σε άλλες περιοχές της Αφρικής. Έχουμε διαφορές σαν παράδειγμα και σε σχέση με τα EPA ε, ξέρουμε ότι η πλειοψηφία των χωρών της περιοχής μας έχουν ήδη υπογράψει μια ενδιάμεση συμφωνία. Ε, μόνο οι κομόρες δεν έχουν υπογράψει τη συμφωνία, αλλά νομίζω ότι θα το κάνουν σύντομα. Νομίζω λοιπόν ότι σε επίπεδο πολιτικό η Επιτροπή του Ινδικού Ωκεανού έχει παίξει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια επίτευξης πολιτικής λύσης στην Μαδαγασκάρη. Δεν έχουμε ολοκληρώσει ε, την προσπάθεια και πάντα εκπλησόμεθα από τις αλλαγές στη Μαδαγασκάρη, αλλά μπορούμε να είμαστε περίπου βέβαιοι ότι η διαδικασία πλέον ε, δεν μπορεί να ακολουθήσει διαφορετική κατεύθυνση και θα, υπάρξει, θα υπάρξουν εκλογές προεδρικές και νομοθετικές ο πρώτος γύρος τον Οκτώβριο και ο δεύτερος τον Δεκέμβριο. Η επίλυση της πολιτικής, ε, του πολιτικού προβλήματος στη Μαδαγασκάρη οφείλεται και στην προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Αφρικανική Ένωση είχε δώσει εντολή στη ΣΑΝΤΕΚ, την ε, Περιφερειακή Συνεργασία των χωρών της Νότιας Αφρικής. Παρ' όλα αυτά, λόγω ακριβώς των στενών σχέσεων που έχουμε με τις χώρες αυτές, και στα πλαίσια της συνεργασίας με τις χώρες του Ινδικού ωκεανού συνεργαστήκαμε, συνεχίσαμε την προσπάθεια έτσι ώστε να υπάρξει επιστροφή στην συνταγματική τάξη στην Μαδαγασκάρη και η, αυτό που θα ονόμαζε η περιφερειακή μας εμπειρογνωμοσύνη μας επέτρεψε να κάνουμε προτάσεις στη Διεθνή Ομάδα Επαφής ιδιαίτερα στην τελευταία συνάντηση στην Άντις ε, οι οποίες προτάσεις πράγματι οδήγησαν στην έβρεση μιας λύσης αποδεκτής και από πλευράς ε, της ε, διεθνούς αν θέλετε κοινότητας αλλά και από πλευράς των ιδίων των κατοίκων της Μαδαγασκάρης. Γιατί φυσικά θα ήταν επικίνδυνο να επιβάλλουμε στους Μαδαγασκαριανούς μια έξοδο από την κρίση η οποία θα μπορούσε να ερμηνευτεί καθιοδήποτε τρόπο σαν μια επιβολή ακριβώς από πλευράς των χωρών της διεθνούς κοινότητας. Οι λύσεις λοιπόν θα πρέπει να δοθούν από τους ίδιους τους ε, κατοίκους της Μαδαγασκάρης. Εμείς θα πρέπει ε, να πιέσουμε και το πετύχαμε αυτό ε, έτσι ώστε τα δικαστήρια και ιδιαίτερα το ανώτατο δικαστήριο της Μαδαγασκάρης να ξαναβρούν την αξιοπιστία τους γιατί αλλιώς θα αντιμετωπίζαμε τεράστια προβλήματα γιατί ακριβώς αυτό το δικαστήριο καλείται να επικυρώσει τα αποτελέσματα των επομένων εκλογών. Και γι' αυτό ζητήσαμε το ανώτατο αυτό δικαστήριο να αναδιαρρυθμιστεί, να υπάρξουν νέα μέλη και με προεδρικό διάταγμα του ε, μεταβατικού προέδρου και έτσι μπορέσαμε να λύσουμε αν θέλετε σε αυτή τη φάση το συγκεκριμένο θέμα. Η σταθερότητα της Μαδαγασκάρης είναι κρισιμότατη για τη σταθερότητα την περιφερειακή. Εμείς ε, οι μικρές χώρες, ε, ε, εμείς στα πλαίσια της συνεργασίας του Ινδικού ωκεανού δεν θα μπορέσουμε να ευημερίσουμε αν η Μαδαγασκάρη δεν πάρει τη θέση που της αξίζει στο σύνολο των εθνών του κόσμου. Είναι ο σιτοβολώνας άλλωστε της περιοχής και παίζει σημαντικό ρόλο όχι μόνο για τις δικές μας χώρες νήσους αλλά και για την Νότια γενικά και την Ανατολική Αφρική. Γι' αυτό λοιπόν οι ανησυχίες μας δεν είναι ακριβώς οι ίδιες με τις χώρες της Υπηρετικής Αφρικής αλλά οι στόχοι θα έλεγα συμπίπτουν με τους στόχους των φίλων. Σας ευχαριστώ για τις παρεμβάσεις σας και για τις απαντήσεις σας. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ. Θα τελειώσουμε λοιπόν τη συνεδρίασή μας σήμερα. Η επόμενη συνάντηση θα γίνει στις 30 Σεπτεμβρίου και στις 3 Οκτωβρίου από τις 9 μέχρι τις 12.30. Σας ευχαριστώ. Καλό απόγευμα σε όλους. Merci messieurs. Oups. Merci beaucoup.